Uh, Συνάδελφοι, να αρχίσουμε την ε, συνεδρίαση. Πριν όμως αρχίσει το σημείο με το οποίο θα αρχίσουμε την συνεδρίασή μας, με δύο λόγια να σας ενημερώσω. Να σας πω, χθε το απόγευμα τι συμφωνήσαμε οι συντονιστές. Όπως γνωρίζετε, συζητήσαμε το περιεχόμενο αυτές της επιστολής για το κατά πόσο είναι κατάλληλη υποψήφη για τη θέση του Επιτρόπου και οπότε αυτή η επιστολή είχε διανεμηθεί σε όλους τους συντονιστές πριν υπογραφή από την Πρόεδρο. Επίσης είπαμε για κάποια άλλα θέματα εκρεμή από την εκτή θητεία, κοινοβουλευτική θητεία και συμφωνήσαμε οι συντονιστές να συζητηθεί σήμερα αυτό το σχέδιο επιστολής από την ε, Επιτροπή. Έχετε λάβει το σχέδιο της επιστολής. Τώρα, όσον αφορά τις αποστολές και την προσωπία, οι πράσινοι πρότειναν να στείλουμε μια αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, να δούμε τι δουλειά θα κάνει εκεί και να μας υποβάλουν τις προτάσεις τους για να καταρρίσουμε το πρόγραμμα. Επίσης έχουμε κάποιες εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας και αποφάσισαν οι συντονιστές να γίνει συζήτηση για το τι θα κάνουμε για το πρόγραμμα που αφορά τι ε, χώρε τη Βαλτική. Και όλα αυτά με την επιφύλαξη του τι θα αποφασιστεί στο μέλλον για, να γίνει τελικά η έκθεση δίας πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό τη Βαλτική. Επίση, είπα στι πολιτικέ ομάδες να κατεβάσουν τι προτάσει του για, για τις υπόλοιπες εκθέσεις δίας πρωτοβουλίας και σα ευχαριστώ που με ακούσατε και τώρα. Αρχίζουμε τη σημερινή μα δουλειά με το πρώτο θέμα τη σημερινή διάταξη. οπότε και ε, θερμά καλωσορίζουμε τη Σουηδική Προεδρία. Θα την εκπροσωπήσει σήμερα <laughs> η κυρία Μοντ, όλο που είναι Υπουργό Επιχειρήσεων και Ενέργεια, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου ε, για την ε, Συνοχή. Και επίση έχουμε και τον κύριο Χέγκλουντ που είναι ε, υπουργό. Πάρα πολύ αξιόλογο και αυτό γιατί μάλλον θα τα λέμε συχνά κατά την Προεδρία. Και θα είστε εσείς και κύριε όταν δεν μπορεί η κυρία Όλαυσον να ε, έρχεται εδώ να μας δει. Οπότε σας παραδίδω αμέσω αμέσως στη σκητάλη για να κάνετε την εισήγησή σας για την Προεδρία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, θα ήθελα να αρχίσω με συγχαρητήρια προς όλους εσάς για την εκλογή σας. Είναι πολύ σημαντική η αποστολή σα και ξέρω βέβαια ότι ορισμένοι από εσά είναι καινούργοι εδώ. Αλλά από την άλλη μεριά είναι πάρα πολύ συναρπαστικό να ασχολείται με το ευρωπαϊκό όραμα, να ανοίγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και εγώ έχω διατελέσει μέλο ε, τη Ρίξτατ, του, του Σουηδικού Κοινοβουλίου και είναι πάρα πολύ σημαντικό το, το έργο που επιτελούμε. Οπότε, καλή επιτυχία ολόκληρο εκ μέρου μα. Επίση, φέρουμε να υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μαζί σα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε. Και έτσι η Προεδρία να σημειώσει πάρα πολλέ επιδόσεις. Είναι δύσκολη η συγκυρία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρίση στο κλίμα, κρίση στην οικονομία. Έχουμε τη διάσκεψη Κοπενχάγη, καινούργιο κοινοβούλιο, καινούργια επιτροπή. Έχουμε πολλά μπροστά μα και γι' αυτό το λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε ούτω ώστε να μπορέσουμε όλε αυτέ τι προκλήσει να τι αντιμετωπίσουμε και αυτό για το καλό τη Ευρώπη. Εσεί, τα μέλη τη Επιτροπή τη Περιφερειακή Πολιτική, θα πρέπει να βοηθήσετε την περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και την πολιτική συνοχή στην Ευρώπη διότι πρόκειται για κάποιες ε, πολιτικές οι οποίες πρόκειται να συμβάλλουν στο να γίνει περισσότερη η ε, ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να έχουμε καλύτερη κοινωνική συνοχή στην Ένωση, γιατί θα πρέπει οι διαφορές, τα χάσματα, τα περιφερειακά να μειωθούν. Και η Ευρώπη, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις. Όπως προείπα, έχουμε την χρηματοοικονομική κρίση, αλλά έχουμε επίσης και αυτού του είδους την οικονομική ύφεση ε, η οποία έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Τα διαποτελέσματα αυτής της κρίσης είναι αισθητά παντού στον κόσμο. Βεβαίω για, για κάποιους η κρίση ήταν χειρότερη από ό,τι για άλλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της τώρα θα πρέπει να δουν πώς θα μπορέσουν να φτάσουν κάποια βιώσιμη ανάπτυξη και πώς θα έχουμε ε, κάποιο είδου ε, ανταγωνιστικότητα, γιατί χρειάζεται να έχουμε καλύτερε επιδόσει στον τομέα τη απασχόληση, αλλά χρειάζεται επίση να έχουμε περισσότερη ευημερία για του πολίτε μα, αλλά και στην Ήπεθρο. Πάρα πολύ σημαντικό επομένω να μπορέσουμε να δούμε πώ θα αποκτήσουμε περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε αυτέ οι διαφορέ θα γεφυρωθούν και δεν θα αυξηθούν διαφορέ μεταξύ των περιφερειών. Παρά το ότι σοβεί αυτή η κρίση δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το ότι θέλουμε να πετύχουμε μακρόπνοια ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να κατευθυνθούν προσπάθειες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε ενωσιακό. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική η πολιτική συνοχή και άρα θα πρέπει να, να ταινίζουμε αυτόν τον τρόπο προ το μέλλον. Και έτσι, έτσι θα έχουμε μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, εποχή που θα ακολουθήσει την κρίση. Ξέρετε, αυτές οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να δημιουργηθεί σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να βλέπουμε μακρόπνο, τόσο ώστε να έχουμε τις καλύτερες συνθήκες όλων των περιβάλλων για τις επιχειρήσεις, διότι ε, σε μια συγκυρία τέτοιων κρίσεων και θα πρέπει να προχωρήσουμε επί τη βάση στρατηγικής που έχουμε χαράξει. Να έχουμε κάποιες στρατηγικές μακρόπονες για τις περιφέρειες και επίση θα πρέπει να απλουστευτεί η διαδικασία λήψη αποφάσεων και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα ταμεία με έναν τρόπο απλούστερο, να μπορέσουμε να επηρεάσουμε περισσότερο τις τοπικές περιφερειακές αρχές και να εκμεταλλευτούμε με πιο πιθανό τρόπο τους αλλά για αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο, θα πρέπει να έχουμε περισσότερο συντονισμό μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών. Θα γνωρίζετε ότι έχουμε κατεβάσει κάποιε προτάσει για να αλλάξουν οι διατάξει που ισχύουν όσον αφορά τα διευθυντικά ταμεία, ώστε να τα απλουστεύσουμε και να είναι πιο εύκολη η εφαρμογή, η υλοποίηση των προγραμμάτων. Πάρα πολύ σημαντικέ αυτέ οι προτάσει. Και όχι μόνο επειδή τώρα έχουμε την, την κρίση, αλλά η Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί για να υλοποιήσει αυτές τις προτάσεις, αυτές τις μεταβολές. Σε επίπεδο ομάδων εργασίας του Συμβουλίου, αυτά αρχίσανε από χθε σαν συζητήσεις και θα πρέπει βέβαια να έχουμε και τη δική σας συνένεση για την υλοποίηση των προτάσεων. Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για την εξέλιξη των συζητήσεων και περιμένουμε να έχουμε μια πάρα πολύ θετική συνεργασία. Τώρα, η απλούστευση της λειτουργίας των διαστικών ταμείων είναι κάτι πάρα πολύ ευκταίο, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η απλούστευση, ιδίως από πλευράς των αποδεκτών των ε, κοινωτικών πόρων. Να δούμε σε τοπικό, σε περιφερειακό επίπεδο τι θα κάνουμε, ε, και επειδή έχω ασχοληθεί με τέτοιου είδου προγράμματα, ξέρω πόσο σημαντική υπόθεση είναι. Χρειάζεται αυτή η απλούστευση για να έχουμε εκλογικευμένη, σωστή χρήση των κοινοτικών πόρων. Τώρα, αυτέ οι συζητήσει για την πολιτική συνοχή είναι παλιά υπόθεση και θα συνεχιστεί η προβληματική. Να σα πω τα σημεία κλειδιά κάτι γνώμη μου, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ πολιτικής συνοχής και στόχων της ε, ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Επιχειρηματικό πνεύμα, καινοτομία, ανάπτυξη, θα τα έχουμε συνεχώς κατά νου, περισσότερες, καλύτερες θέσεις απασχόλησης και κοινωνική κάλυψη. Η διαστατική προσέγγιση μέχρι τώρα έχει πετύχει και έχει βοηθήσει να βελτιώσουμε την εκτέλεση των προγραμμάτων. Επίσης, ξέρουμε καλύτερα τους πόρους μας και καταβάλλονται προσπάθειες να υπάρχει συνεχώς μια αξιολόγηση ούτως ώστε να έχουμε εγγύηση μακρόπνοης ε, επιτυχίας των προγραμμάτων και επίσης να έχουμε σε ευρία βάση συνεργασία, συνεργασία σε κάθε επίπεδο και έτσι να έχουμε καλύτερη εκτέλεση των προγραμμάτων. Οι πόροι των διαστικών ταμείων θα πρέπει να συνεχίσουν να επικεντρώνονται σε αυτούς που περισσότερο τους χρειάζονται. Όλοι θα πρέπει να είναι στέση, να ζουν αξιοπρεπώς, να έχουν κάποια παιδεία, κατάρτιση, να υλοποιούν τους στόχους της φιλοδοξίας τους παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι απλά θέμα αλληλεγγύης. Έτσι εξασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Περισσότερη ανάπτυξη στις πιο αδύναμες περιοχές και αυτό προς όφελος όλης της Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, εδαφική συνεργασία, όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε κατά νου, διασυνοριακή συνεργασία, συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, γιατί όλα αυτά αποτελούν προσθέμενη αξία για όλη την Ένωση. Πρέπει να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα μέτωπα. Η κάθε περιφέρεια έχει τις δικές της ε, αρετές που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Στο νότο έχουμε το καλό κλίμα, ε, τουρισμό, αλλά και στον βορρά πολλά μπορεί να γίνουν. Να, ε, όπως αυτά τα ξενοδοχεία που φτιάξανε από πάγο. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι ζουν σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να δώσουν να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Γι' αυτό σας λέω ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στις ε, επιτόπου εμπειρίες και έτσι να χαράσετε σχετική πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πρόκειται να διοργανώσουμε στην Κυρούνα, στη Βόρεια Σουηδία, μία διάσκεψη. Διαλέξαμε αυτό το μέρος με μεγάλη προσοχή. Διότι προσθέσεις μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η περιοχή είναι παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε. Η Κυρούνα είναι πολύ βόρεια, πολύ μακριά. Πάνω πάνω στη Σουηδία είναι αεροκατοικημένη περιοχή, πρόκειται για κάποιο... Εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ορυκτά, εκεί κατοικεί η φυλή των Σάμι. Εκεί υπάρχει ένα τέτοιο ξενοδοχείο από πάγο. Έχουμε εγκαταστάσεις ε, ε, Παρακολούθηση του διαστήματο. Επομένω δεν πρόκειται μόνο για μια περιοχή που είναι το χειμώνα σκοτεινή με πολύ χιόνι. Η μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι θα τολμήσει να έρθει Και πάνω η Ντανότα Χούμνερ για να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα τόσο σημαντικά. Και προσοχή, όποιος τολμήσει να έρθει εκεί γιατί είναι πάρα πολύ κρύα εκεί πέρα, ήδη από τώρα. Επομένω, εκεί θα δούμε πώ μπορεί κανεί να εκμεταλλευτεί τι επιτόπου δυνατότητε και πώ μπορεί κανεί να θεμελιώσει την ανάπτυξη, πώ μπορεί κανεί να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που με με καλύτερο τρόπο. Επίση, να δούμε ποια είναι η στρατηγική που θα εκμεταλλευτεί τι πρώτε ύλε, που και αυτό βοηθά την ε, οικονομία. Εμεί χαιρετίζουμε αυτή την ε, ενωσιακή πρωτοβουλία είναι ό,τι καλύτερο τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη και θέσει αποσχόληση. Τώρα, όσον αφορά την ανάπτυξη των πόλεων, σε σχέση με την πολιτική εδαφικής συνοχής. Και εδώ θα πρέπει να επεξεργαστούμε κάποια κριτήρια. Πώς θα πετύχουμε εδώ περισσότερη ανάπτυξη. Πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τη μεταβολή του κλίματος, όσον αφορά την ένταξη, γιατί η συνοχή είναι σημαντική και όσον αφορά τις μακροοικονομικές στρατηγικές. Και εδώ μπαίνει η στρατηγική μας για την Βαλτική. Είμαστε βέβαιοι ότι αν έχουμε μια στρατηγική διασυνοριακή, τότε έχουμε τις προϋποθέσεις αντιμετώπισης των στόχων μας. Αλλαγή του κλίματος, περιβάλλον, αντιμετώπιση της κρίσης. Η δε πρόταση θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική ένταξη. Και έτσι θα ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά, θα έχουμε καλύτερες επενδύσεις στις υποδομές και η Βαλτική θα πλησιάσει ούτως υπήν την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνουν επενδύσεις επίσης έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και στην ανάπτυξη. Αυτή η στρατηγική δεν προϋποθέτει περισσότερους πόρους. Αντίθετα, θα εκμεταλλευτούμε τα υπάρχοντα προγράμματα. Θα τα τρέξουμε πιο αποτελεσματικά και θα έχουμε καλύτερο συντονισμό και συνεργασία. Να γίνει δηλαδή συντονισμός των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και όλα αυτά τα συζητήσουμε αρχά Οκτωβρίου. Θα τα συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή σα αλλά και η Προεδρία από κοντά θα παρακολουθεί τι εξελίξεις και έτσι ελπίζουμε ότι κατά τον τρόπο θα μπορέσουμε τις απόψει σα να τις ε, περιλάβουμε ε, στις δικές μας προτάσεις. Όλες αυτές τις προτάσεις που θα έχουμε για την στρατηγική μας. Παγκοσμιοποίηση, αλλαγή του κλίματος, ενέργεια, δημογραφικές μεταβολές. Όλα αυτά είναι προκλήσεις. Και βεβαίως τα διορθωτικά ταμεία ήδη καλύπτουν αυτούς τους στόχους, αλλά εμεί θα πρέπει να δούμε στο μέλλον πώς αυτές οι επενδύσεις θα συνδεθούν με την συνοχή, την κοινωνική και οικονομική. Γιατί πάντα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θέλουμε οικονομική βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον. Το θέλουμε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον. Και θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να συνδυαστεί η οικονομία με την βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρειάζονται. Χρειάζεται αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, αλλά χρειάζονται και καινοτομίες στην τεχνολογία. Και έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, αλλά ταυτόχρονα να μειώσουμε το ίχνος το οποίο αφήνουμε στον πλανήτη από τη χρήση της ενέργειας. Ήδη έχει εικονοφραστεί ε, ποια κονδύλια θα για μια πράσινη οικονομία και είναι κάτι που θα συνεργαστεί μετά το 2013. Αυτή η μετάβαση προς μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον είναι για μας προτεραιότητα. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να τα βλέπουμε σαν συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Ήδη έχει αρχίσει αυτή, αυτός ο μετασχηματισμός παντού στην Ευρώπη και αν όχι όλοι, πάρα πολλοί ηγέτες Ευρωπαίοι είναι πρωτοπόροι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχουν συνειδητοποιήσει ότι εάν εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρει αυτή η αλλαγή προς μια φιλική στο περιβάλλον οικονομία, τότε θα έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα για πολύ καιρό στο μέλλον. Έχει μοναδική ευκαιρία η Ευρώπη. προκειμένου το ώστε να αποκτήσει πρωτοπόρο ρόλο να αποκτήσει το πλεονέκτημα. Αυτό το μήνυμα θέλει να στείλει η Σουηδική Προεδρία. Για αυτή την πολιτική έχουμε πολλά εργαλεία στη γεωργία, στις ΜΜΕ, στην καινοτομία, στη συνοχή, σε όλες, όλες αυτές οι πολιτικές είναι παραδείγματα εύστοχα του πώς είναι δυνατόν κανείς να πάει προς μια τέτοια αλλαγή προς μια πράσινη οικονομία. Και εσείς εδώ, στο Κοινοβούλιο και στην Περιφερειακή Επιτροπή συγκεκριμένα, έχετε ένα τέτοιο ρόλο στη, διαμόρφωση του μέλλοντος για την Ευρώπη. Πολλοί στη σημερινή συγκυρία χρειάζονται ε, μια υπεύθυνη πολιτική ηγεσία, πρωτοπορία, ούτω ώστε να ενδυναμωθεί η Ευρώπη, να έχουν περισσότερες θέσεις εργασίας και έτσι όλος ο κόσμος να έχει εμπιστοσύνη στο μέλλον. Είμαι βεβαίω ότι θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά, θα ακούσουμε τις θετικές σας ε, εμπειρίες και προτάσεις και έτσι πιστεύω θα βγούμε από αυτή την κρίση πιο ενισχυμένη, πιο δυνατή. Σα ευχαριστώ την προσοχή σα. Ευχαριστώ να απαντήσω τι τυχόν ερωτήσει που έχετε και να ακούσω τι άλλο έχετε να μου πείτε για να το λάβω υπόψη και να το διαβιβάσω αρμοδίω στην Προεδρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για την εισαγωγή σας που δείχνει ότι τα μεγάλα μελήματά σας στην πολιτική, την περιφερειακή και την πολιτική συνοχή είναι ίδια με τα δικά μας. Επομένως, τους επόμενους μήνες μπορούμε να συνεργαστούμε, να συνεργαστούμε. Μιλήσατε για την Εταφική συνοχή, για το μέλλον αυτής της πολιτικής, για την ατζέντα της Θησαβόνας, που είναι πολύ σημαντική για την πολιτική μας. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσει η συζήτηση. Η Υπουργός περιμένει και ερωτήσεις, αλλά και σχόλια. Θα ήθελα να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Ας ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Χάρηκα ιδιαίτερα που η Σουηδική Προεδρία θέλει να θέσει στο προσκήνιο την στρατηγική για την Βαλτική και το αναφέρω αυτό γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πολιτική με τη Ρωσία και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η πολιτική για την Βαλτική. Ίσως θα μπορούσατε να μας κάνετε κάποιες παραπάνω παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις αυτές με τα τρίτα κράτη. Έχω όμως και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Δυστυχώς όπως κάθε καλοκαίρι είχαμε μεγάλες πυρκαγιές. Το συζητήσαμε και χθε στην Επιτροπή. Και για μένα το ερώτημα που ανακύπτει είναι πάντα το εξή. Έχουμε το Ταμείο αλληλεγγύη το Συμβούλιο, το οποίο υπάρχει εδώ και καιρό. Σκοπεύει η Σουηδική Προεδρία να το θέσει σε κίνηση και να επιχειρήσει να απλοποιήσει τον κανονισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο προκειμένου να είναι πολύ πιο ευέλικτη η αντίδρασή μας σε περίπτωση που πλήττονται κάποια τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από φυσικές καταστροφές. Δεύτερη ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι η στρατηγική για τη Βαλτική αποτελεί εδαφική στρατηγική, αλλά θα ήθελα να ακούσω και δύο λόγια για το πώς θέλετε να προωθήσετε την εδαφική συνοχή. Υπάρχει η πράσινη βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τοποθετήθηκε σχετικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να συζητήσουμε και να συνεχίσουμε τις σχετικές συζητήσεις. Θα ήθελα όμως και κάποιες παρατηρήσεις ε, εκ μέρους σας. Uh, θα ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις ε, πρώτα και μετά θα απαντήσει ο Υπουργός. Γιάνν Ολμπρίχτ. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Μιλώ συντονιστής του ΕΛΚΑ στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στην Προεδρία και στο Συμβούλιο. Άκουσα τη θέση της Προεδρίας, της Σουηδικής Προεδρίας αλλά από διαφορετικές προεδρίες ακούσαμε διαφορετικές απόψεις για το τι είναι η πολιτική συνοχής. Άκουσα το λόγο σας σήμερα και άκουσα διαφορετικά στοιχεία από αυτά που έχω ακούσει στο παρελθόν. Υπουργέ, μιλήσατε για τα στοιχεία της ε, Ατζέντα Λισαβόνας στην πολιτική συνοχής. Υποτίθεται για να προωθηθεί η καινοτομία, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε στις πιο ισχυρές και δυνατές περιοχές. Αλλά η πολιτική αυτή είναι θέμα ίσων ευκαιριών ε, και τις δυνατότητες που δίνουμε στις ε, ασθενέστερες ε, περιφέρειες να πιάσουν τις πιο ισχυρές. Δεν θα πρέπει να κοιτάξουμε το δεύτερο στόχο της πολιτικής συνοχής. Ε, γιατί μπορεί να προωθήσει πολύ την ασύγκληση. Ακούω διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές απόψεις. Η Σουδική Προεδρία θα προωθήσει την απλούστευση. Είναι σημαντικό η πολιτική συνοχή να εμπλουτιστεί, ούτω ώστε να υπάρχουν ωφέλη για όλη την κοινότητα, ε, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο για κάποιες περιοχές. Μία ερώτηση προς το Συμβούλιο παίρνουμε ανεπίσημες πληροφορίες για κάποιες αντιφάσεις που υπάρχουν στο... και αντιρρήσεις που υπάρχουν στο Συμβούλιο για την απλούστευση του κανονισμού εν ώψη της τρέχουσας κρίσης. Θα ήθελα να ρωτήσω την Υπουργό να μας πει ποια είναι η διάθεση στο Συμβούλιο, ποια είναι η τάση σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στον κανονισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να επηρεάσουν την, ευρωπαϊκή, την κοινωνική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Άλλη μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις για τα θέματα που θα προωθήσει η Προεδρία σας. Θα ήθελα να αναφέρω ότι με τη Γαλλία και την Τσεχία είχαμε θαυμάσια συνεργασία, αλλά και με εσά όταν προετοιμάσαμε το μακρόπνο πρόγραμμά σας. Ακόμη και οι τοπικές αρχές ενεπλάκησαν, γιατί η εμπλοκή των τοπικών αρχών είναι πολύ σημαντικό να θέσουν και αυτές ε, τους στόχους, τις προτεραιότητές τους για το μακροπρόθεσμο πρόγραμμά σας. Εσείς μιλήσατε για το σημαντικό ρόλο των πόλεων ε, των Δήμων και Κοινοτήτων ε, στη λήψη των αποφάσεων. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Πώς θα βελτιώσετε και θα τις ενσωματώσετε καλύτερα στις όλες τις στρατηγικές. Πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί πιστεύω ότι με την εμπλοκή αυτή θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τα κονδύλια. Ε, για τις περιφερειακές πολιτικές μίλησατε για τις προτεραιότητες, παράδειγμα το χάρη στη Βαλτική. Τι πιστεύετε για αντίστοιχες περιφερειακές στρατηγικές, παραδείγματο χάρη τη στρατηγική του Δούναβη, ας πούμε, των περιοχών του Δούναβη ή άλλων περιοχών. Δεν υπάρχουν επικαλύψεις ανάμεσα αυτές τις περιφερειακές στρατηγικές και, σε, και στην πολιτική συνοχής. Θα ήθελα τώρα ο Υπουργός να δώσει τις απαντήσεις της. Ευχαριστώ για τις απόψεις αλλά και τις ερωτήσεις. Ας ξεκινήσω με τη στρατηγική της Βαλτικής, που ήταν η πρώτη και τελευταία ερώτηση που άκουσα. Νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος αυτός για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα εργαλεία ε, για να συνεργαστούμε καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και περιμένω πραγματικά με υπομονησία να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γιατί όλοι εστιάζουν στο στόχο της καλής συνεργασίας. Όταν συνεργαζόμαστε με εταίρους, πρέπει να, είμαστε ανοιχτοί στις ιδέες τους. Η συνεργασία δεν πρέπει να είναι κλειστή στη φύση της, πρέπει να είναι ανοιχτή. Ξέρω ότι γίνονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή για διάφορα προγράμματα με τρίτες χώρες και αυτό είναι πολύ καλό και σημαντικό. Αλλά πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό όταν μιλάμε για την ε, περιοχή της Βαλτικής ή του Δούναβη, ας πούμε, να εντοπίσουμε για ποιο λόγο θέλουμε να συνεργαστούμε και να το συζητήσουμε. Θα πρέπει από την αρχή να εστιάσουμε, ειδικά στην αρχή, στα σημαντικά στοιχεία, στις σημαντικές προτεραιότητες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια πλατιά συνεργασία και μια πλατιά συζήτηση. Από πλευράς της Σουηδικής Κυβέρνησης θα ήθελα να πω ότι έχουμε εμπλέξει πολλά υπουργεία, πολλούς υπαλλήλους, πολλά τμήματα της κοινωνίας μας σε αυτή την ε, συνεργασία για τη Βαλτική. Και επιμερίζουμε τις ευθύνες μεταξύ διαφορετικών Υπουργείων και Φορέων, ούτω ώστε να υπάρχει πραγματική λογοδοσία αργότερα από όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπλακεί στη διαδικασία. Επομένως, νομίζω ότι είναι πολύ καλό και πραγματικά μας εμπνέει αυτή η συνεργασία και ο τρόπος που προγραμματίζεται για τη Βαλτική. Το θέμα δεν είναι μόνο πολιτική συνοχή. Δεν προσπαθούμε μόνο να συνδέσουμε τη Βαλτική και τις χώρες Βαλτικής με την πολιτική συνοχή. Χθε ήμουν στην Επιτροπή Ήτρε και εκεί συζητούσαμε πώς θα μπορούσαμε να, συνδέσουμε σε ό,τι αφορά τα θέματα ενέργειας τις χώρες της Βαλτικής, τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Παραδείγματος χάρη με νέα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε λοιπόν τέτοιες χώρες, όμορες χώρες. Το θέμα είναι να έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα, όχι μόνο προγράμματα τα οποία θα είναι ατελέσφορα. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης, χαιρόμαστε που τα πράγματα επιτέλους αρχίζουν να κουνιούνται, γιατί επί... μακρόν είχαμε βαλτώσει. Τώρα προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά πιο αποτελεσματικά. Η Προεδρία μας θα εστιάσει σε αυτό το θέμα και οι επόμενες Προεδρίες. Και όπως είπα και στην εισαγωγή μου, αν βρίσκεστε από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, αν είσαστε αποδέκτης της βοήθειας, ξέρετε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι τα πράγματα να δουλεύουν αποτελεσματικά. Επομένως, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει όλοι να το ψάξουμε, να δούμε πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα πράγματα καλύτερα. Τώρα για την εδαφική συνεργασία, οι συζητήσεις που θα κάνουμε στην Κυρίνα ε, θα είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η εδαφική συνεργασία. Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει προστιθέμενη αξία σε αυτό. Αν δείτε ότι διαφορετικές περιφέρειες Ευρώπης έχουν διαφορετικές συνθήκες ε, και τις αθροίσετε όλες αυτές τις ε, συνθήκες και προϋποθέσεις, βλέπετε τις, ε, τη δύναμή μας, αλλά και τις αδυναμίες μας πρέπει να δουλεύουμε με τις άλλες περιφερειές αλλά με πρακτικό τρόπο. Και αν κοιτάξετε την κρίση που, έχουμε αυτή τη στιγμή, που περνάμε αυτή τη στιγμή στη Σουηδία αλλά και σε άλλες χώρες, αυτό που κάναμε στη Σουηδία είναι να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική συνοχή και τις διάφορες εταιρικέ σχέσεις που έχουμε εδραιώσει, ούτω ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα για να βοηθήσουμε αυτούς που χάσαν τη δουλειά τους καταρχήν. και να βοηθήσουμε το, τον κόσμο με απτό, με πρακτικό τρόπο. Πολλές από αυτές τις δομές, πολλοί από αυτούς τους φορείς ε, ε απέδειξαν την αξία τους με πρακτικό τρόπο. Όλα αυτά τα ταμεία, όλα αυτούς τους φορείς θέλουμε να τους ε, καταστήσουμε πιο αποτελεσματικούς, λιγότερο γραφειοκρατικούς. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μελλοντική πολιτική συνοχής. Ξέρω ότι διαφορετικέ χώρε βλέπουν το μέλλον αυτή τη πολιτική με διαφορετικό τρόπο. Και δεν είναι μυστικό να σα πω ότι και διαφορετικά πολιτικά κόμματα έχουν τελείω διαφορετικέ απόψει για αυτά τα ταμεία και τα κονδύλια τη πολιτική συνοχή. Το θέμα είναι να βρούμε μια κοινή οδό που θα πρέπει και οι 27 χώρε να την υποστηρίξουν και φυσικά να συμφωνήσουν. Ούτω ώστε η πολιτική συνοχή να είναι ενεργή, να δίνει αποτελέσματα. Αν οι πολιτικές αυτές καταστούν πιο αποτελεσματικές και συνδεθούν με τους στόχους της Λισαβόνας, μπορούμε περαιτέρω να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά τους. Α, στο μέλλον όμως, οι πιο αδύναμες περιοχές είναι αυτές που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και εκεί πρέπει να πάνε οι περισσότεροι πόροι. Χώρες όπως η Σουηδία θα χρησιμοποιήσουν τους εθνικούς τους πόρους για να βοηθήσουν τις δικές τους αδύναμες περιοχές, γιατί αυτές είναι ήδη ισχυρές χώρες. Νομίζω όμως ότι αυτή η συζήτηση, ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει. Μια καλή συζήτηση. Όσο πιο αποτελεσματική γίνεται η πολιτική συνοχή, όσο πιο καλή είναι η διάρθρωσή τη με άλλε πολιτικέ, με άλλου φορεί, παραδείγματο χάρη με το χτίσιμο μια πράσινη οικονομία, τόσο πιο χρήσιμα θα είναι αυτά τα κονδύλια, τόσο πιο χρήσιμα θα είναι αυτά τα ταμεία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εντοπίσουμε τι προτεραιότητε τη πολιτική συνοχή. Τώρα, για το αν υπάρχουν διαφωνίες στο Συμβούλιο για το θέμα της απλούστευσης. Κοιτάξτε, δεν έχουμε βγάλει και τα μαχαίρια. Αλλά ο καθένα έχει τι δικέ του ιδέε για την απλούστευση. Τώρα, από τι ιδέε και τι υποδείξει πρέπει να περάσουμε σε συγκεκριμένε αποφάσει. Και συχνά έχουμε την ε, τάση να προτάσουμε τι δικέ μα εθνικέ ιδέε και πολιτικέ. Όντω γίνεται μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το πώ θα απλουστεύσουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του κανόνε. Προσπαθούμε να συμφωνήσουμε για να έχουμε τα καλύτερα τα αποτελέσματα. Και εδώ θέλω τη βοήθειά σας, ούτω ώστε να εμπλουτιστεί η συζήτηση, να ακούσουν και άλλες ιδέες για το πώς θα απλουστεύσουμε καλύτερα τη διαδικασία. Τώρα, για τις πόλεις, τις κοινότητες, τους δήμους, πώς μπορούμε να τι εμπλέξουμε στην διαδικασία με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η έχω εγώ εμπειρία γιατί βρέθηκα από την άλλη μεριά του τραπεζιού. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ε, στις πόλεις, σε δήμους, κοινότητες που έχουν όρεξη να ανακατευτούν. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένοι από μια τέτοια δουλειά, από μια τέτοια προσπάθεια. Και η μεγάλη πρόκληση για μας είναι ε, οι μικρέ επιχειρήσει, οι οργανώσει των γυναικών, οι οι μικρές, οι μικροί φορείς να εμπλακούν στην όλη προσπάθεια. Εμείς ως πολιτικοί θα πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ε, μέσα σε μια πλατιά βάση να πούν την άποψή τους να ακούσουμε συγκεκριμένες ιδέες και να εμπνευστούμε από αυτές. Επομένως, η ευρεία εταιρική σχέση είναι πολύ σημαντική. Θα ήθελα να τονίσω την ευκαιρία που έχουν και οι επιχειρήσεις. Συχνά οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή να εμπλακούν σε αυτή τη συζήτηση, να πούν την άποψή τους. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την ανάπτυξη στο μέλλον, πρέπει να καταλάβουμε πώς θα γίνουν περισσότεροι επιχειρηματίες, πώς θα ανοίξουν περισσότερες δουλειές, πώς θα υπάρχουν, υπάρχουν περισσότερες εταιρικές σχέσεις, πώς θα μπουν περισσότεροι άνθρωποι στην αγορά εργασίας. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Υπουργέ Όλεψον. Η πολιτική συνοχή έχει καταφέρει στο παρελθόν να συμβάλλει στην σταθεροποίηση διαφόρων περιφερειών και στην ανάπτυξή τους. Και τώρα βρισκόμαστε ενώπιον δύο μεγάλων ερωτημάτων. Καταρχάς, πώς η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αξιολογηθεί, πώς μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα και κατά δεύτερον, ε, ανακύπτει το ερώτημα εν, το μέσο της κρίσης κατά πόσο αναπτύχθηκαν καλές δομές σε περιφέρειες οι οποίες χρειάζονται βοήθεια και θα ήθελα να θέσω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Καταρχάς, ποια είναι η θέση της Σουηδικής Προεδρίας σε ό,τι αφορά το θέμα της αξιολόγησης, της μέτρησης των αποτελεσμάτων ως τώρα της, συνοχής, ε, της πολιτικής συνοχής. Και κατά δεύτερον, έχετε ενδείξεις που σας κάνουν να πιστεύετε ότι κάποιες ισχυρές περιοχές πλέον θα καταστούν περιοχές ε, αποδέκτες ε, βοήθειας. Αναφέρατε επίσης το θέμα της επιτάχυνσης της ε, καταβολής των κονδυλίων και η σχετική πρόταση της Κομισιόν μας έχει ήδη διατεθεί. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν πρόκειται για ένα μέτρο που αποσκοπεί σε συγκεκριμένους στόχους σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτή την ανάληψη πιστώσεων. Έχει το Συμβούλιο μια επισκόπηση για το ποιες χώρες επί του παρόντος δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πιστοτικές υπηρεσίες, άρα εξαρτώνται 100% από την καταβολή αυτών των κονδυλίων, γιατί είμαι βέβαιος ότι δεν είναι 100% η εξάρτηση για όλες τις χώρες και ότι μπορεί να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και με άλλους τρόπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλφόνση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Υπουργέ, ευχαριστώ. Μιλώ εξ, ονόματι, εξ ονόματος των Πράσινων. Ακούσαμε τα λόγια σας, τα εκτιμήσαμε εμπολής, ειδικά αυτά που είπατε σε ό,τι αφορά την πρόθεσή σας να καλλιεργήσετε τις διαφορετικές κουλτούρες. Εγώ είμαι από την Κορσική και με ενδιαφέρει πάρα πολύ οι διάφορες κουλτούρες της Ευρώπης να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της πολιτιστικής πολυμορφίας που είναι η όψη και η σφραγίδα της Ευρώπης. Επίσης, είπατε ότι θέλετε να προωθήσετε την ανάπτυξη των ασθενών περιφερειών και η Ευρώπη θα στηριχθεί ε, στο δυναμικό αυτών των περιφερειών και στην ε, διασυνοριακή συνεργασία. Δείξατε με το παράδειγμα της Βαλτικής ε, πώς μεγάλες, μεγάλοι χώροι ιστορικοί και οικολογικοί προσεγγίζονται μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας. Φαντάζομαι ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η Μεσόγειος. Εγώ σαν Γκόρσος εκπλήσωμαι όταν βλέπω πόσο αδιάφορες είναι οι πολιτικές ανάμεσα ε, για την, ε, τις ανταλλαγές ανάμεσα στους ανθρώπους. Ε, Παραδείγματο χάρη, εμείς είμαστε δίπλα στην ε, Σαρδινία και όταν τελειώνει η τουριστική περιοχή ξεχνάμε ότι υπάρχουν οι άλλοι, οι Σάρδοι. Η Προεδρία σας σε αυτό το τομέα δεσμεύεται ίσως να προωθήσει βαθιές μεταρρυθμίσεις ούτως ώστε οι διασυνοριακές πολιτικές να πάνε πιο μακριά, πιο βαθιά για να υπάρξουν περισσότερες ε, ανταλλαγές μεταξύ των λαών που ανήκουν στον ίδιο χώρο, στην ίδια φυσική λεκάνη. Ευχαριστώ κύριε Σκότμαν, σε ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο στοιχεία να ρωτήσω. Καταρχάς, ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας σε ό,τι αφορά την πολιτική για την αλλαγή του κλίματος και για την πολιτική της συνοχής. Την κλασική πριν τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα για την πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, ε, πιστεύω ότι είναι πιο ισχυρό το πρόγραμμα για την ε, κλιματική αλλαγή, αλλά πώς θα είναι η διάδραση μεταξύ των πολιτικών αυτών, πώς θα συνδέσετε αυτά. Αυτό είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση, μια προκλητική μάλλον ερώτηση. Ε, η κατάσταση στο Συμβούλιο θύχτηκε. Και να σας πω, όταν βρισκόμαστε σε κρίση, όταν τα κράτη-μέλη καλούνται να καταπολεμήσουν την ενεργεία, προσπαθούμε να επενδύουμε στις ε, υποδομές. Αλλά θα τεθεί και θέμα ανταγωνισμού. Γιατί δεν είναι το θέμα μόνο να βελτιωθούν οι υποδομές, αλλά και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα όταν θα εκδηλωθεί η κρίση. Και αν διαρκέσει πολύ αυτή η διαδικασία, το πρόβλημα θα είναι ακόμα πιο οξύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Τελευταία συνάδελφος που ζητάει το λόγο, Ρίκα. Α, βλέπω ότι υπάρχει όμως και άλλος ομιλητής που ζητάει το λόγο, άρα να δώσω τον λόγο στην Υπουργό πρώτο. Πρώτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις αυτές που μου θέσατε σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχής και την αξιολόγησή της. Είναι αυτονόητο, εννοείται. Η πολιτική συνοχής, αν θέλουμε να την υπερασπιστούμε, θα πρέπει να αποδείξουμε ποια είναι και τα αποτελέσματά της. Και τα τελευταία χρόνια μιλάμε για το συνδυασμό της πολιτικής συνοχής με άλλες στρατηγικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό για τον Ευρωπαίο πολίτη να αναφέρεται στα προγράμματα τι γίνεται και με τον προϋπολογισμό. Θα πρέπει ασφαλώς να κάνουμε ένα απολογισμό του τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Και επίσης να δούμε πότε θα πρέπει οι δράσεις να αναλαμβάνονται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο ή περιφερειακό επίπεδο. Δεν μπορούν όλα να χρηματοδοτούνται σε κινητικό επίπεδο. Θα πρέπει και οι περιφέρειες να συμμετέχουν. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αξιολογήσουμε τώρα για την επόμενη περίοδο. Υπάρχουν όμως δυνατότητες αξιολόγησης. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να σημειώσω, σε ό,τι αφορά και την τελευταία ερώτηση, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι η πολιτική συνοχή αποτελεί ένα μόνο τμήμα. Υπάρχουν και τα σχέδια ανάκαμψης, υπάρχουν και τα εθνικά σχέδια, τα εθνικά προγράμματα, τα μέτρα για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Γιατί φυσικά θα πρέπει να διευκολυνθεί και η κυκλοφορία της ρευστότητα στις τράπεζες. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να είναι αλληλοσυνδεόμενα σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρξει αυτή η επιτάχυνση της ε, καταβολής των κονδυλίων. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα η συζήτηση για την συγχρηματοδότηση και για ποιο τμήμα θα πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση προς την κατεύθυνση αυτή και θα πρέπει να υπάρχει και συνεισφορά των κρατών, γιατί αυτό θα συνεπάγεται και μια ευθύνη για τα προγράμματα αυτά, γιατί καταλαβαίνω, μένω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό για τα κράτη-μέλη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Όταν χρησιμοποιούμε φορολογικούς πόρους, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και εθνικοί περιφερειακοί πόροι. Πρόκειται για μια συζήτηση φυσικά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και γενικά διατυπώνονται πάρα πολλέ διαφορετικέ απόψει ε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό ο πολιτισμός στην Ευρώπη να ενισχυθεί. γιατί τώρα τονίσαμε την πολιτική για τη Βαλτική, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αποτελεί ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα πιο αποτελεσματικής διαμόρφωσης των εργασιών μας. Και θεωρώ ότι τα όσα συμβαίνουν για την πολιτική για το Δούναβη, για τη Μεσόγειο, παραβρέθηκα το καλοκαίρι στο Μιλάνο και κάναμε σχετικές συζητήσεις, πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα εντυπωσιάστηκα από όσα συμβαίνουν στην περιοχή της Μεσογείου. Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή. Νομίζω ότι θα πρέπει να ελέγξουμε νέε μεθόδου για τι εργασίε μα, προκειμένου να μάθει και ο ένα από τον άλλον, να διδαχθούμε ο ένα από τον άλλον. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική για το κλίμα, την πολιτική για την συνοχή και κατά πόσο υπάρχει μια εγγενή αντίφαση. αντίφαση. Όχι, αντιθέτω θεωρώ. Η Σουηδία θεωρεί ότι εδώ και τώρα που έχουμε την οικονομική κρίση, εδώ και τώρα πρέπει να οικοδομήσουμε ένα νέο όραμα για την Ευρώπη. Πού είναι λοιπόν οι νέες δυνατότητες για την Ευρώπη, οι νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Ξέρουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει στον τομέα της αλλαγής του κλίματος. Θα πρέπει να περιορίσουμε τις εκπομπές μας. Και αυτό τι σημαίνει θα πρέπει να αναπτυχθούν καινούρια επιχειρηματικά προγράμματα, νέες πηγές ε, ενέργειας, νέοι τρόποι μεταφορών, επικοινωνία, τεχνολογία επικοινωνίας. Υπάρχουν τόσο μεγάλες ευκαιρίες στον τομέα αυτό που δεν αρκεί να είμαστε από τους καλύτερους. Όχι, θα πρέπει να είμαστε οι καλύτεροι και νομίζω ότι πραγματικά ε, η πολιτική για το κλίμα αποτελεί μια εξαιρετική βάση για την ανάπτυξη αυτή. Και να σας πω ότι από τις επαφές μου με τη ΣΥΠΑ, με την Κίνα, διαπιστώνω ότι και οι άλλες ε, πλευρές κάνουν μεγάλες επενδύσεις. Και είδα χθε στην Επιτροπή Βιομηχανίας, συζητήσαμε για διάφορα προγράμματα, διαπιστώνουμε ότι και οι άλλοι λοιπόν κάνουν μεγάλες επενδύσεις. Και εμείς λοιπόν θα πρέπει να επενδύσουμε επιπρόσθετα. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ όντως να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της βιώσιμης οικονομίας. Να δημιουργηθεί μια νέα βιομηχανική ανάπτυξη, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Υπό την έννοια αυτή δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ της κοινοτομίας και της ε, πολιτικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος, όταν μιλώ για περιβάλλον και για την ανάπτυξη της οικονομίας, πρόκειται πραγματικά για έναν τέτοιο διτό στόχο. Και στο πλαίσιο αυτό θα είναι σημαντική και πολιτική συνοχή για να πετύχουμε το αποτέλεσμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη Υπουργέ, σα ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις ε, θέσει σας και τις φιλοδοξίες που μας παρουσιάσατε για την περιφερειακή πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό ότι τονίζετε ακριβώς στα πλαίσια της Προεδρίας σας την περιφερειακή πολιτική. Ακούσαμε πολλά και σημαντικά ερωτήματα. Θα ήθελα όμως να συζητήσω την στρατηγική με την Βαλτική, για τη Βαλτική και στο πώς σχετίζεται με την περιφερειακή πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντική η στρατηγική για τη Βαλτική, για τις χώρες αυτές. Και όπως ακούσαμε, είναι σημαντικό να συνδεθεί με ευρωπαϊκά θέματα, αλλά κοιτώντας και τα παράκτια κράτη της Βαλτικής περιοχής, αυτό που μας ε, κάνει εντύπωση είναι ότι δεν πρόκειται για μια πολιτική η οποία ωφελεί μόνο τις πόλεις, αλλά και την ύπεθρο στις χώρες αυτές. Προκειμένου και οι χώρες αυτές να αναπτύξουν τη δική τους περιφερειακή πολιτική. Εσείς, κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας, πώς σκοπεύετε να ενεργήσετε προκειμένου και άλλες πόλεις, πέρα από τις παράκτιες πόλεις, να αποκτήσουν ένα σύνδεσμο με την πολιτική για την Βαλτική θάλασσα. Γιατί πραγματικά είναι σημαντικό να τεθεί επί ευρεία βάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Σέμπερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τα λόγια της ε, Υπουργού για την πράσινη οικονομία. Ένα βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι οι τιμές για τη συμβατική ενέργεια είναι μάλλον χαμηλές. Άρα η δομή των τιμών που διαμορφώνεται στην αγορά θα είναι κάτι το οποίο δύσκολα θα μπορούμε να ξεφύγουμε. Ενώ για παράλληλα η αιωλική ενέργεια είναι μάλλον ακριβή. Άρα ήθελα να σας ρωτήσω, σκοπεύετε να παρέμβετε σε τιμολογιακό επίπεδο προκειμένου να ενισχύσετε την πράσινη ενέργεια. Θέλετε να εισάγετε πιλωτικά προγράμματα. Γιατί φυσικά πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του πετρελαίου και του αερίου. Ένα δεύτερο ερώτημα. Ένα βασικό θέμα το οποίο εμπλέκεται σε πολλά ευρωπαϊκά θέματα είναι η γραφειοκρατία. Τι συζητιέται λοιπόν σήμερα στο Συμβούλιο για την μείωση της γραφειοκρατίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους αυστηρούς ελέγχους των προγραμμάτων. Έχετε μήπως κάποιες καινούργιες ιδέες για να υπάρξει κάποια πιο χαλαρή διαχείριση σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Και τρίτο ερώτημα, ποιους δείκτες συζητάει το Συμβούλιο αναφορικά με τον ορισμό των περιφερειών. Μιλάμε για το κατακεφαλή εισόδημα. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς εξελίσσονται οι συζητήσεις από αυτή την άποψη. Ο τελευταίος ομιλητής, Γιώργος Ματούλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Μία μικρή ερώτηση έχω, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Είμαι Ρουμάνος, από τη Δυτική Ρουμανία. Και θα ήθελα να μιλήσω για τις ε, μικρές επιχειρήσεις, αλλά και για τις όχι και τόσο μικρές. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση αυτής της πρόσβασης στα κοινωτικά κονδύλια. Έχω πολλά παραδείγματα να σας δώσω. Μερικές φορές οι επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη πολυεθνικές συχνά, έχουν καταθέσει προγράμματα για να λάβουν χρηματοδότηση και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. 1.700 νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν στο εσωτερικό μιας επιχείρησης σε αυτή εδώ την κρίσιμη περίοδο, την περίοδο κρίσης πήγαν σε ανθρώπους ε, από μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες. Αυτές οι επιχειρήσεις ε, ζητούν την περίοδο της κρίσης μέσα για να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει να πλουστευτεί η διαδικασία αυτή. αν δεν υπάρχουν γρήγορα, αν δεν γίνονται γρήγορα αυτές οι χρηματοδοτήσεις, αυτά τα project δεν θα καταλήξουν. Και οι επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να τα καταφέρουν όπως όπως με διαφορετικό τρόπο. Ειδικά όταν πρόκειται για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να δοθούν αυτά τα κονδύλια. Θα πρέπει αυτά τα θέματα να εξεταστούν στο εσωτερικό του Συμβουλίου και να απλουστευτούν οι διαδικασίες. Ευχαριστώ. Ακόμα μία ερώτηση, τελευταία. Ζητώ συγγνώμη, καμιά φορά σας μπερδεύω, δεν βλέπω τα καρτελάκια σας. Υπουργέ, Είμαι από μια χώρα της Βαλτικής. Και σας συγχαίρω που η στρατηγική της Βαλτικής είναι μια από τις προτεραιότητές σας. Αλλά όταν ήμασταν στο Στρασβούργο, πολλοί συνάδελφοι έθεσαν το εξής ερώτημα. Ε, είναι μεν προτεραιότητα η στρατηγική αυτή, αλλά δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι. Πώς γίνεται αυτό, ρώτησαν οι συνάδελφοι. Θα μπορούσατε να μας διαβεβαιώσετε ότι στον επόμενο προϋπολογισμό θα υπάρξουν αρκετοί πόροι για τη στρατηγική της Βαλτικής. Γιατί χωρίς πόρους η στρατηγική αυτή θα παραμείνει κενό γράμμα. Είμαι Εστονή, που είναι η μικρότερη χώρα, η Εστονία είναι η μικρότερη χώρα της Βαλτικής. Μιλήσατε πάρα πολύ για συνεργασία και ανάπτυξη. Τι μπορείτε να πείτε στην Εστονία. Έχουμε 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους, 1,3 εκατομμύρια και το 50% από αυτούς είναι άνεργοι. Είναι μια εθνική καταστροφή. Το 50% του εργατικού δυναμικού μας είναι άνεργοι. Έχετε κάποιες προτάσεις. Τελείωσαν τα σχόλια και οι ερωτήσεις. Θα ήθελα τώρα η Υπουργό να κάνει τις τελευταίες δηλώσεις της και να απαντήσει τις τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, ακόμα μια φορά. Χαίρομαι που τόσοι πολλοί από εσά ενδιαφέρονται για τη στρατηγική της, Λισαβ... της και θέσαν τόσες ερωτήσεις. Θεωρώ ότι αυτό μαρτυρά το ενδιαφέρον όλων μας για να συνεργαστούμε. Είναι μια νέα εξέλιξη στην πολιτική, λένε όλοι, και αυτό μπορεί να είναι για όλους. Ακούστηκε μια ερώτηση για το πώ μπορούν να υποφεληθούν από αυτή την πολιτική και άλλε περιοχέ των χωρών και όχι μόνο οι παράκτιε περιοχέ. Νομίζω ότι οι κυβερνήσει και οι εθνικές οργανώσεις θα πρέπει να το δουν αυτό το θέμα. Γιατί η, Βαλτική, η στρατηγική της Βαλτικής δεν είναι μόνο για τι παράκτιε περιοχέ, είναι για όλη την περιοχή τη Βαλτική. Επομένω, οι εθνικέ κυβερνήσει και οι εθνικέ οργανώσει θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι εμπλέκουν και τις υπόλοιπες περιοχές των χωρών της Βαλτικής, όχι μόνο τις παραθαλάσσιες, τις παράκτιες. Καλό είναι που θέσατε αυτό το ερώτημα. Από την εμπειρία που έχω μέχρι τούδε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όλη η περιοχή να είναι τμήμα της στρατηγικής της Βαλτικής. Να πάω τώρα στο τελευταίο ερώτημα που τέθηκε από την Εστονή κυρία. Αν δούμε τώρα τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή, η στρατηγική της Βαλτικής, μην ξεχνάτε δεν ε, σημαίνει νέος προπολογισμό. Σημαίνει απλώς χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε ήδη και τα καθιστούμε πιο αποτελεσματικά. Κατά την άποψή μου, αλλά κα, κατά την άποψη πολλών άλλων, το θέμα είναι πώς μπορούμε να εμπλέξουμε περισσότερους ανθρώπους, να δημιουργηθούν νέες καινοτομίες, ε, νέες ιδέες και τελικά νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτό τι σημαίνει. Μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών, ούτως ώστε να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Περισσότερες ευκαιρίες στις αγορές. Στην κυβέρνησή μου είμαι υπεύθυνη για την βιομηχανία και, το, και τις επιχειρήσεις. Και η συνεργασία που έχω μεταξύ της Σουηδίας και των υπόλοιπων χωρών της Βαλτικής σε αυτό το τομέα είναι πολύτιμη. Αλλά μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για να ενδυναμώσουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. για να αυξήσουμε, να παραπλασιάσουμε τι ευκαιρίε που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει για να βγουν στην αγορά, στη μεγάλη αγορά, πέρα από την εθνική αγορά. Χθε συζητήσαμε στην Επιτροπή Ήτρε το θέμα τη απλούστευση των κανόνων. Και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα κοιτάζει αυτό το θέμα. Αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό το θέμα. Πώ θα μειώσουμε την γραφειοκρατία. Είναι καθήκον όλων μα να βοηθήσουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει να ανθίσουν γιατί έτσι παράγεται πλούτο στην Ευρώπη, γιατί έτσι δημιουργείται ανάπτυξη στην Ευρώπη. Παραδείγματο χάρη, ηλιακή ενέργεια, αιωλική ενέργεια. Α, ήταν μια άλλη ερώτηση. Και πώ μπορούμε να παίξουμε με τι τιμέ, Αν θέλουμε να εισαγάγουμε νέε μοντέρνε βιώσιμε ενέργειε σε μια εισαγωγική φάση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολλαπλού τρόπου, πολλαπλέ ε, ενεργειακέ τεχνολογίε. Στην Ευρώπη έχουμε διάφορα συστήματα. Παραδείγματο χάρη στην ε, Σουηδία, έχουμε ένα σύστημα που βασίζεται στην αγορά, που λειτουργεί καλά για να προωθήσουμε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ε, με αυτόν τον τρόπο ε, πολλαπλασιάζονται οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια όταν βασιζόμαστε στην αγορά. Άλλε χώρε έχουν άλλο σύστημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε ε, νέες μορφές ενέργειας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα πρέπει να παγιωθούν σε μια κατάσταση. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη για, την, ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παραδείγματο χάρη η Ιδανία, η Γερμανία και η Σουηδία έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της αιωληνικής ενέργειας. Είμαστε οι καλύτεροι μαθητές. Τα πράγματα έχουν ε, αλλάξει τελείω σε σχέση με 20 χρόνια πίσω. Αν κοιτάξετε 20 χρόνια πριν δεν είχε καμία σχέση. Δεν είχαμε καθόλου αιωλική ενέργεια. Είναι μια τεράστια, ένα τεράστιο δυναμικό αυτό της αιωλικής ενέργειας. Ε, θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε εδώ δεν είναι απλώς ότι σώζουμε το περιβάλλον, αλλά προωθούμε και ένα νέο βιομηχανικό κλάδο ε, που τον χρειάζεται η Ευρώπη για να δημιουργήσει και απασχόληση κτλ. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό. Ένα άλλο τρόπο για να υποστηρίξουμε την ε, οικονομία μα είναι η καινοτομία, η έρευνα και η ανάπτυξη. Έχουμε διάφορα προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν, ε, υπάρχει το σχέδιο ανάκαμψης που μιλάει για τις επενδύσεις. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε για να σπρώξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που συμβαίνει στη Σουηδία τουλάχιστον είναι ότι πολλές τοπικές εταιρείε και πολλές πόλεις δίνουν τα χέρια σε συνεργατικές μορφές ε, για να προωθήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, πιστεύουμε ότι αυτό ε, συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο. Για να περάσουμε σε ανανεώσιμες και να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έπειτα, για τα θέματα του ελέγχου. Εφόσον χρησιμοποιούμε τα λεφτά του φορολογούμενου, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Από την άλλη, όμως, τα πράγματα που αφορούν τον έλεγχο των προγραμμάτων πρέπει να πλουστευτούν. Ε, νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο συχνά ρίχνουμε το φταίξιμο στην Ευρώπη. Κάθε φορά που υπάρχουν προβλήματα φταίει η Ευρώπη. Κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο φταίει η Ευρώπη. Εγώ στη Σουηδία ως Υπουργό έχω την ευθύνη να εξασφαλίσω ότι τα δικά μας προγράμματα είναι αποτελεσματικά. Αλλά νομίζω ότι και στην Ευρώπη έχουμε ευθύνη ούτως ώστε να απλουστεύσουμε τα πράγματα. Γιατί όπως ανέφερε και ένας βουλευτής, είναι πολύ σημαντικό οι πόροι που έχουμε προβλέψει να φτάσουν στα χέρια αυτών που προβλεπόταν να φτάσουν. Ε, μία κουβέντα για την κρατική υποστήριξη. Συζητήσαμε τις ανησυχίες της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως ξέρετε, μέσα στο 2009 πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία. Μια ισορροπία μεταξύ μιας μορφής υποστήριξης που κινδυνεύει να γίνει μακροπρόθεσμη και των υγιών συνθήκων ανταγωνισμού. Μακροπρόθεσμα υποστηρίζουμε το ανοιχτό και ελεύθερο εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων. Ίσως όμως βραχυπρόθεσμα να χρειαστεί να υπάρξει και κρατική υποστήριξη. Και ο ίδιος ο τομέας λέει ότι μόλις θα επανέλθει σε υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού θα ξεφύγει, θα αποκοπεί από αυτή την υποστήριξη, την κρατική υποστήριξη. Νομίζω ότι απάντησα σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Θα ήθελα συμπερασματικά να πω και κάτι άλλο. Και δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Αλλά συμπερασματικά θέλω να σας πω ότι πραγματικά μου είναι πολύτιμη η συνεισφορά σας και τα σχόλιά σας. Και δεδομένου ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι μπορεί. Αντιμετωπίζει την κρίση. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να παραμείνουμε στις δάφνες μας. Θα πρέπει να κονίσουμε τα εργαλεία μας για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο μέλλον. Έχουμε πάρα πολλές δεξιότητες στην Ευρώπη. Πάρα πολλά προσόντα, πάρα πολλές δυνατότητες. Νομίζω ότι μπορούμε να τι αξιοποιήσουμε. Ήταν καλό που έγινε αυτή η πρώτη συζήτηση μαζί σα. Και αν δεν έρχομαι κάθε φορά εδώ, δεν θα έρχομαι στο μέλλον κάθε φορά εδώ, σημαίνει ότι έχω πολλές άλλες υποχρεώσεις, υπουργικές υποχρεώσεις και δεν θα μπορώ κάθε φορά να είμαι παρούσα, αλλά θα παρακολουθώ τα τεκτενόμενα. Σας ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες ιδέες σας, για τη συνεισφορά σας και ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εξ όλων των συναδέλφων στην αίθουσα αυτή. Πρέπει να σας πω ότι ε, πραγματικά εκτιμούμε τη δεσμευσή σας στην πολιτική σας ατζέντα, η οποία είναι και πολύ φιλόδοξη για τους επόμενους μήνες. Όπως είπατε και στην αρχή, ως υπουργό ε, καλύπτεται πάρα πολλού τομεί. Αυτό όμω είναι και πολύ θετικό γιατί σας δίνει μια ενιαία, αν θέλετε, προσέγγιση σε πολλά θέματα. Και όπως ξέρετε, όλα τα θεσμικά όργανα έχουν τη δική τους ατζέντα. Και εδώ στο Κοινοβούλιο από την Επιτροπή μας περιμένει ο κόσμος να κάνει ό,τι μπορεί το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας για να ενισχύσει την κατάσταση. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Και γι' αυτό λοιπόν εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δέσμευσή σας. Ελπίζω και τους επόμενους μήνες και καταρχάς τον Οκτώβριο να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να πετύχουμε από κοινού πιο πολλά. Σας ευχαριστώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δύο λεπτά διάλειμμα. Να χαιρετήσουμε τον Υπουργό και θα περάσουμε στο 10 της ημερήσιας διάταξης. Uh, Σωρά. Can we start, can we continue? Να συνεχίσουμε. More time to, for all the points. So I would like... Για να μην καθυστερήσουμε και με τα υπόλοιπα σημεία. It's back. Καθίστε. Move to point number 10. I would like to... Να περάσουμε στο 10. να σας ενημερώσω, το ανέφερα και χθες, ότι λάβαμε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μία επιστολή, η οποία απεστάλλει σε όλους τους Προέδρους των Επιτροπών αναφορικά με τα εκκρεμή ζητήματα από την έκτη νομοθετική περίοδο και σε ό,τι αφορά επίσης τις ε, προτεραιότητες για την τρέχουσα θητεία. Μας ζητάει λοιπόν ο Πρόεδρος την επιστολή μέχρι 9 Σεπτεμβρίου να χορηγήσουμε τις πληροφορίες από την ε, Επιτροπή μας σε ό,τι αφορά τους κανόνες 114, 54 και 119 ενδεχόμενες τροπολογίες δηλαδή που θα θέλαμε να υποβάλουμε. Για να ανταποκριθούμε λοιπόν σε αυτό το αίτημα του Προέδρου, η Γραμματεία προετοίμασε μια επιστολή η οποία αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αναφορικά με τα εκκρεμή ζητήματα, όπου έχουμε και υποχρέωση να απαντήσουμε. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο τμήμα του σχεδίου της επιστολής μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να το αποστείλουμε. Και το δεύτερο τμήμα απαρτίζεται από τις πολιτικές προτεραιότητες που θα μπορούσαν να προσθεθούν αν θέλετε στο πρώτο τμήμα της επιστολής αλλά αυτό μπορούμε και να το στείλουμε αργότερα μπορούμε και να το στείλουμε και καθόλου αν αυτό θέλουμε. Το σχέδιο λοιπόν αυτής της επιστολής συζητήθηκε χτες ε, στα πλαίσια της συνάντησης των συντονιστών, τροποποιήθηκε και από τις προτάσεις των συναδέλφων των Πρασίνων, της ΓΚΟΕ και του ΕΛΚ. Προσθέσαμε λοιπόν τις τροπολογίες αυτές και η τραποποιημένη αυτή επιστολή σας απεστάλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χτες το βράδυ θα σας το μοιράσουμε κιόλας για να το έχετε μπροστά σας να σας πω ότι το πρώτο τμήμα της επιστολής δεν ε, απασχόλησε ιδιαίτερα τους συντονιστές νομίζω ότι ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης το μόνο εκρεμές ζήτημα είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο δεν είναι όμως αμφιλεγόμενο ως θέμα. Το δεύτερο θέμα μας απασχολεί, το δεύτερο τμήμα για τις προκλήσεις. Να σας πω ότι η δική μου πρόταση θα ήταν να αποστείλουμε και τα δύο τμήματα της επιστολής προς τον Πρόεδρο. Αλλά φυσικά, αν θέλουμε κάτι να αλλάξουμε, κάτι να προσθέσουμε, να κοιτάξουμε το δεύτερο τμήμα της επιστολής. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά. Ελπίζω να γίνει και μια εσβάθων συζήτηση στο άμεσο μέλλον. Να κάνουμε λοιπόν μια πρώτη συζήτηση, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και για το δεύτερο τμήμα, για να αποστείλουμε το σύνολο της επιστολής. Άρα, να συζητήσουμε λοιπόν τώρα το δεύτερο τμήμα της επιστολής. Γιατί εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε κάποια αλλαγή να γίνει ή αν θέλουμε να παραμείνει η επιστολή ως έχει. Άρα, να ρωτήσω τώρα τους βουλευτές αν έχουν κάποια συγκεκριμένα σχόλια. Η Κωνσταντσα Κρέιλ, ευχαριστώ πάρα πολύ Ντανούτα. Δύο σημεία ήθελα να θίξω, τα οποία έθιξα και χτες στην ακρόαση με τον Επίτροπο και σήμερα στην Προεδρία. Το Ταμείο Αλληλεγγύης, από ό,τι κατάλαβα, χρειάζεται περαιτέρω δραστηριοποίηση εκ μέρους του Συμβουλίου. Αλλά είναι σαφές ότι το Συμβούλιο δεν επιθυμεί να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα πιο έντονα, πιο οξύ έναν διατύπωση στην επιστολή αυτή, γιατί δεν είναι δυνατόν να βγούμε και να πούμε στις περιφέρειες ότι το συζητήσαμε στο Κοινοβούλιο, αλλά το Συμβούλιο κάνει πίσω γιατί δεν είναι δυνατόν τα 27 κράτη-μέλη να συμφωνήσουν επί μιας ε, ενιαίας διαδικασίας. Δεν νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο μπορούμε να αποδεχτούμε κάτι τέτοιο. Δεύτερο στοιχείο. Εξ όσων άκουσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από τη, τα σημαντικά σημεία προτεραιότητας ε, της θητείας αυτής, την προετοιμασία δηλαδή των νέων χρηματοοικονομικών προοπτικών μετά το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν σχεδιάζει να συστήσει ομάδα εργασίας και στην ομάδα εργασίας αυτής ε, εκπροσωπούνται όλα τα θεσμικά όργανα η ΕΟΚΕ, η Επιτροπή των Περιφερειών, το Συμβούλιο, η Κομισιόν, όλοι εκεί συμμετέχουν, μόνο το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει. Και μετά ακούμε δηλαδή ότι ο Επίτροπος θέλει να ακούσει τις ε, απόψεις μας. Ε, δεν μας αρκεί αυτό. Ως Επιτροπή πραγματικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να συμφωνήσουμε, να απαιτήσουμε μία θέση, μία έντρα σε αυτή την Επιτροπή είμαστε πώς να το κάνουμε. Οι εκλεγμένοι των όλων των ευρωπαϊκών χωρών με δημοκρατικό τρόπο. Και ίσως θα έπρεπε να το αναφέρουμε και στην επιστολή. Ή να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο τέλο πάντων να διατυπώσουμε με σαφήνεια αυτή τη θέση μας. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Για το Ταμείο Αλληλεγγύης θέλω να σας πω ότι υπάρχει. Ίσως θέλετε να αναφερθεί αυτό πολύ πιο έντονα. Τι αλλαγή ακριβώς θέλετε. Θέλετε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία του Ταμείου Αλληλεγγύης, έτσι. Πολύ ωραία. Για τα υπόλοιπα δεν υπάρχει πρόβλημα. Πολύ ωραία. Άλλα σχόλια. Κύριος Αλφόνς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτο σημείο. Θέλω να επανέλθω σε ένα σχόλιο που υπήρχε στην αρχική επιστολή και που δεν υπάρχει πια. Την παρακολούθηση των διαδικασιών και των μέτρων κατά της κρίσης. Νομίζω ότι το συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα και συμφωνήσαμε. Έπειτα, μετά από αυτά που είπε και η προλαλήσασα, η ομάδα μας θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία διαλόγου μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν όταν εκπονούνται προτάσεις για τη μελλοντική πολιτική συνοχής. Γιατί πραγματικά πρέπει να υπάρχουν ανταλλαγέ απόψε μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Πραγματικέ ανταλλαγέ. Γι' αυτό προτείνουμε αυτή η φάση τη πρώτερη διαβούλευση να αναφέρεται στην επιστολή. Να ζητήσουμε κάτι τέτοιο ρητά, λοιπόν. Απ' τη μία θέλουμε να παρακολουθήσουμε αυτά τα μέτρα κατά της κρίσης. Αυτό θα μπει στο δεύτερο τμήμα και από την άλλη θέλετε αυτό, τη συνεργασία. Εντάξει. Άλλα σχόλια. Κύριος Όρο. Yes. Ευχαριστώ. Και εγώ προφανώς συμφωνώ με την επιστολή. Το είπα και χθε στη συνεδρία των συντονιστών. Διερωτώ όμως, μήπως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο έντονα για μια νέα πολιτική. Γι' αυτή δεν μιλούσαμε προηγουμένως, με την Υπουργό. Αυτή η νέα πολιτική στρέφεται προς την πράσινη οικονομία, προς τα νεώσιμες πηγές ενέργειας. Φυσικά υπάρχει μια απαρχή αυτού του πράγματος στην πρόταση που κάνουν οι πράσινοι. Αλλά νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας, κυρίως ημών που είμαστε στην, ε, πολιτική, στην ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, να τα πούμε αυτά τα πράγματα πιο σαφώς. Είναι ευθύνη μας. Μπορείτε να είσαστε πιο συγκεκριμένος Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι χρειαζόμαστε μια συζήτηση για τη μελλοντική πολιτική και θα την κάνουμε αυτή η συζήτηση. Είναι ένα από τα μείζωνα καθήκοντά μας. Υπάρχει αυτή η τελεία για τις διαπραγματεύσεις για το νομοθετικό πακέτο και την προετοιμασία του νομοθετικού πακέτου. Υπάρχει αυτή η τελεία σας στην επιστολή. Αλλά αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, θα έλεγα να πούμε ρητά ότι πρέπει να συζητηθεί το μέλλον αυτής της πολιτικής. Καλή ιδέα. Θα το βάλουμε αυτό το σημείο. Γιατί ίσως το έχουμε αναφέρει, αλλά με τρόπο πολύ τυπικό. Ε, ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ περισσότερο από τις διαπραγματεύσεις ε, του νομοθετικού πακέτου. Πρέπει να δώσουμε πραγματογνωμοσύνη, πρέπει να συμμετάσχουμε σε όλες τις συζητήσεις, κάτι παραπάνω δηλαδή από αυτό που αναφέρουμε τώρα εδώ με εντελώς τυπικό τρόπο. Άλμπριχτ. έχω να προτείνω μια αλλαγή τεχνικού χαρακτήρα. Εκεί στο δεύτερο μέρος έχουμε τρία διαφορετικά στοιχεία. Το ένα Είχε που λέει ότι δημιουργείται συντάσει στο Συμβούλιο και θα πρέπει κανεί να προσδοκά τέτοιε συγκρούσει και εντάσει και στο Συμβούλιο. Είναι πρόβλημα τη απλούστευση των κανόνων όσον αφορά τα διαρκτικά ταμεία τώρα για του ισχύοντε τρέχοντε κανονισμού. Άρα θα πρέπει αυτό να το ενοποιήσουμε. Για, για το πρόγραμμα ανάκαμψη και λοιπά και όλα μαζί να τα βάλουμε. Και το άλλο το οποίο μόλι τώρα μα ανέφερε η πρόεδρο είναι το ότι θα πρέπει να συζητήσουμε την μέλουσα πολιτική συνοχή. Κάθε αυτή. Και μετά τι, τι, τις του νομοθετικού πακέτου. Και το πρόβλημα τη εδαφική συνοχή. Και το τρίτο είναι η συζήτηση για τη στρατηγική, για την καταπολέμηση των ε, θεομηνιών και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, αυτό σας τονίζω. Θα πρέπει το πρώτο κομμάτι να, να το, χωρίσουμε. Οι ισχύοντες κανονισμοί, ε, πολιτική, πακέτο, τα, τα τρία στοιχεία. Πρόεδρος. Καλά. Να μιλήσετε με την γραμματεία, να το κανονίσετε. Έχετε κάτι άλλο να πείτε. Θα προφτάσουμε, δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει. Τέλο πάντων, θα ελπίζουμε να προλάβουμε και να σα στείλουμε την επιστολή. Και έτσι να μπορέσουμε έγκαιρα να το έχουμε έτοιμο για να το στείλουμε στον κύριο Μπουζέκ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει εδώ κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ή περιμένουμε ένα πεντάλεπτο για να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν να έρθει πιο γρήγορα ο συνάδελφος της Κομισιόν. Τι, τι θέλετε. Εντάξει, δύο, λεφτάκια. Να δω αν ο κύριος Σάνικ μπορεί να έρθει. Για να δούμε, έρχεται είναι στο δρόμο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 Uh, είναι Είναι στο αυτοκινητό του και έρχεται, άρα σε ένα τεταρτάκι θα είναι εδώ. Οπότε να διακόψουμε για αυτό το τεταρτάκι, αν θέλετε να το κάνουμε έτσι. Να ξαναρχίσουμε σε ένα τέταρτο. Σε ένα τέταρτο. Άρα 11 τέταρτο. Τι και Υπότιτλοι Authorwave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 Να ξαναρχίσουμε, συνάδελφοι. Για τους συναδέλφους που έρχονται για πρώτη φορά εδώ στους ευρωβουλευτές ή πρώτη φορά στην Επιτροπή των Περιφερειών θέλω να σας πω ότι ζητήσαμε να έρθει εδώ Γενικός Διευθυντής για την ε, Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ο, ο ομολογός μας με τον οποίο συνεργαζόμαστε σε επίπεδο κομισιών. Πριν του δώσω τον λόγο, υπενθυμίζω ότι τον Ιούλιο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αυτόν τον κανονισμό για πλούστευση, κρίση. Δεν υπήρξε ο χρόνος να συζητηθεί, αλλά ε, ζητήσαμε εμείς μάλλον αλλά χωρίς να μπορέσουμε να το συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα για σήμερα το συζητάμε αυτό πρώτη φορά όσον αφορά την κατανομή των κειμένων ανά εισηγητή. Είπαμε θα είναι για το ΕΛΚ, ε, για τον... Ε, για, ε, κ. εδώ για το ΕΛΚ και να δούμε ποιος θα είναι από τους ε, σοσιαλιστές. Και να, επομένως ο κύριος Γενικός Διευθυντής που θα μας πει πώς έχουν τα πράγματα. Πέστε μας επίπεδο Κομισιόν αλλά και Συμβουλίου. Κύριε Άνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, πρώτα πρώτα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε σήμερα. Αυτή είναι μια πρώτη αλλά πάρα πολύ σημαντική συζήτηση που θα γίνει. Και πέραν του θέματος που σήμερα θα συζητήσουμε, θέλω να σας πω ότι είμαι στη διάθεσή σας, εάν θέλετε να συζητήσουμε άλλα θέματα κατόπιν των προσφάτων εκλογών, οπότε και ανανεώθηκε η εντολή σας. Πρέπει να σας ε, πω ότι δεν μπορώ παρά να ευχηθώ καλή επιτυχία. Επίσης, θερμότατες ευχές προς εσάς κύριε Πρόεδρε. Τώρα έχετε καθήκοντα πάρα πολύ συναρπαστικά. Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε τους επόμενους μήνες ε, και χρόνια, όχι μόνο για την κρίση, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική μας στο μέλλον και κυρίως μετά το 2013. Ήδη σε πολλά κρατημέρια έχει αρχίσει ε, η επεξεργασία αυτού της φάσης για να δούμε πώς θα δώσουμε μαζί σάρκα και οστά σε αυτή την συνεργασία. Επομένως, μας περιμένουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα επόμενα χρόνια. Αυτής, ε, η, αυτή η Επιτροπή είναι ο βασικός εταίρος της δικής μας Γενικής Διεύθυνσης. Φυσικά παρακολουθούμε και την Επιτροπή Προϋπολογισμού, την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, αλλά αυτή εδώ η Επιτροπή θεωρούμε ότι είναι ο βασικός μας εταίρος, ο βασικός μας συνομιλητής και με τον προηγούμενο Επίτροπο κάναμε πολλές προσπάθειες για να βελτιώσουμε τις σχέσεις με την Επιτροπή σας και να υπάρξει μεταξύ μας μια πραγματική εταιρική σχέση. Και ο νέος Επίτροπός μου θα ήθελε να κινηθούμε πάλι προς αυτή την κατεύθυνση στο παρελθόν και μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν η Επιτροπή σας ε, μας βοήθησε πολύ και μας υποστήριξε πολύ. Και πραγματικά είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη της Επιτροπής σας. Υποστήριξη απέναντι στις ε, περσινές μας προτάσεις του περσινού Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου χρειάστηκε να τις περάσουμε βιαστικά για να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν. Τότε το Κοινοβούλιο επανέλαβε πολλές φορές ε, την ανησυχία του ότι η διαχείριση των ταμείων και ότι η διαχείριση των πολιτικών μας, η εφαρμογή των πολιτικών μας ε, επιτόπου θα πρέπει να απλουστευτεί. Αυτός είναι ένας στόχος τον οποίο απόλυτα συμμεριζόμαστε. <coughs> Και είμαι πραγματικά ευτυχής ε, που σήμερα σας παρουσιάζω τη δουλειά που κάνουμε σε αυτό το τομέα. Φυσικά γνωρίζουμε τις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την επιθυμία να επιλακίσει σε όλες τις ε, πρωτοβουλίες για όλες τις πολιτικές από την αρχή. Και δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ από πλευράς μας για να γίνει πραγματικότητα αυτό. Θα ήθελα να πω δύο λόγια τώρα για τις προτάσεις μας και για την, ε, κυρίως για τις προτάσεις για την απλούστευση που κάνουμε στο πλαίσιο αυτό κρίσης που βρισκό, βρισκόμαστε. Ίσως θα θυμάστε το δεύτερο εξάμεινο του 2008 όπου ξεκινήσαμε μια νέα εμπειρία με τους ε, συναδέλφους ε, στα νέα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των πολιτικών επιτόπου και για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν με τους κανόνες των πολιτικών. Ξεκινήσαμε λοιπόν στο δεύτερο εξάμεινο του 2008 να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε την περίοδο 2007-2013, την τρέχουσα περίοδο, να απλουστεύσουμε τους κανόνες των πολιτικών, ειδικά στις πιο επίγουσες περιπτώσεις, εκεί όπου χρήζουν εκεί όπου χρήζει απλούστευσης. Παραδείγματος χάρη στα προγράμματα που αποδίδουν, που είναι κερδοφόρα. Γιατί είχαμε πάρα πολλά άχθη, πολλά βάρη, ακόμη και, και στα πιο αργά προγράμματα, στα, πιο, στα λιγότερα επίγοντα. Είχαμε πει λοιπόν ότι θα εξαιρέσουμε τα μικρότερα προγράμματα, ακόμη και αν ε, αποδίδουν ε, κέρδη από αυτούς τους ε, περίπλοκους κανόνες. Κάτι που από διοικητικής πλευράς πραγματικά ήταν πολύ εποφελές. Ενώ ταυτόχρονα σε επίπεδο παρακολούθησης και σε επίπεδο δαπανών κρατήσαμε τους βασικούς μας κανόνες. Δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη τα χάσματα των κερδών και για το βασικό όγκο των εξόδων παραμείναμε ε, πιστοί στους παλιούς κανόνες. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η αλλαγή ήταν ανακούφιση για τα κράτη-μέλη, για τις διοικήσεις των κρατών μελών κτλ. Στα πλαίσια του πρώτου πακέτου για την κρίση της Κομισιόν, το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2008, κάναμε και ένα δεύτερο γύρο προτάσεων για να βελτιώσουμε τους κανονισμούς μας και να απλουστεύσουμε τους κανόνες. Το κάναμε αυτό μετά από ε, πολλές επαφές με εμπειρογνώμονες στα κράτη-μέλη, εμπειρογνώμονες που δουλεύουν επί τόπου και που έχουν την εμπειρία και το κάναμε μετά από συμβουλές που μας δώσαν και τα μέλη της Επιτροπής σας. Σας λάβαμε υπόψη, υπόψη μας γιατί πραγματικά εκπροσωπείτε αυτούς που δουλεύουν επί τόπου και όπου προωθούν την περιφερειακή ανάπτυξη και που είναι οι βασικοί αποδέκτες και δικαιούχοι αυτής της ανάπτυξης. Αυτές οι προτάσεις που κάναμε στο τέλος του 2008, στο μεταξύ υιοθετήθηκαν. Αλλάξαμε κατά συνέπεια και τους εφαρμοστικούς κανόνες που υπάρχουν στον κανονισμό της Επιτροπής και χρησιμοποίησαμε αυτή την ευκαιρία για να διατρέξουμε τον κανονισμό της Κομισιόν για να δούμε τι άλλο μπορεί να πλουστευτεί. Και εκεί, σε συμφωνία με τους εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη, κάναμε κάποιες περαιτέρω πλουστεύσεις και καταλήξαμε σε ένα τρίτο πακέτο πλουστεύσεων. Αυτό είναι το πακέτο που έχουμε τώρα ενώπιόν μας. Σε ό,τι αφορά την οργάνωση και το πώς δουλεύουμε, ε, εξακολουθούμε να δουλεύω μια μικρή διευθύνουσα της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζιο για την απλούστευση. Όλες οι υπηρεσίες συνεργάζονται και εξετάζουμε τι μπορεί να απλουστευτεί για να έχουμε καλύτερη επαφή με αυτό που συμβαίνει επί τόπου στις περιφέρειες. Ζητάμε από τους εμπειρογνώμονες των περιοχών που ασχολούνται με την διαχείριση και τον έλεγχο των πολιτικών μας, ζητάμε από αυτούς να έρθουν στις Βρυξέλλες και να συζητήσουν μαζί μας το κάναμε στα πλαίσια μιας ομάδας όπου είχαμε και εμπειρογνώμονε από τα κράτη-μέλη. Και είχαμε και πολλέ πολλές όμως επαφές με περιφερειακές οργανώσεις. Με εμπειρογνώμονες από το περιφερειακό επίπεδο. Όλες αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν σε αυτό το τρίτο πακέτο που είναι μπροστά μας σήμερα. Οδήγησαν σε αλλαγές ή σε προτινόμενες αλλαγές στους κανόνες. Αυτό το τρίτο πακέτο, αν υιοθετηθεί, αυτό θα σημαίνει ότι, ότι θα ξανααναθεωρήσουμε τους εφαρμοστικούς κανόνες για να τους υιοθετήσουμε παράλληλα με τις αλλαγές στον κανονισμό. Και ελπίζω ότι αν δουλέψουμε σκληρά μαζί, μέχρι το τέλος του 2009 θα μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για την περίοδο του 2007-2013 και το τι μπορεί να γίνει μέσα σε αυτή την τρέχουσα περίοδο. Ε, νομίζω ότι αυτά αρκούν για αυτή την περίοδο, εκτός και να ανακαλύψουμε κάτι όλος διόλου λάθος. Γιατί πρέπει να σταματήσουμε τις αλλαγές για αυτή την περίοδο 2007-2013. Για τον απλό λόγο ότι Τώρα έχουμε περάσει τη φάση της εφαρμογής των πολιτικών. Και νομίζω ότι κατά την εμπειρία μας, με βάση την εμπειρία μας, ε, είναι λάθος να αλλάζουμε τους κανόνες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δημιουργεί μεγάλη σύγχυση, γιατί είμαστε ήδη στο τρίτο πακέτο. Είμαστε χρονικώς ποσοριακοί για ό,τι μπορούμε να κάνουμε, πόσες αλλαγές μπορούμε να προωθήσουμε. Θεωρούμε τώρα ότι η πολιτική από το καλοκαίρι και μετά αρχίζει πραγματικά να πιάνει ρίζες. Και λαμβάνουμε πολλές αιτήσει για επιστροφή χρημάτων από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό είμαι πραγματικά πιο αισιόδοξο για την εφαρμογή της πολιτικής τώρα, πολύ πιο αισιόδοξο από ότι ήμουν στις αρχές του 2009. Τώρα ας περάσουμε στις προτάσεις. Είναι μια πρόταση που εντάσσεται στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Και φυσικά ο στόχος της πρότασης, κατά συνέπεια, είναι διτός. Καταρχάς, να απλουστεύσουμε τις πολιτικές μας, προφανώς. Βεβαίως, θέλουμε να βγάλουμε, να πετάξουμε κανόνες που είναι περιττοί, που δημιουργούν σύγχυση, περιπλοκές. Αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις περιπλοκές και τις δυσκολίες, μπορούμε, μπορούμε να τις αποφύγουμε. Θέλουμε όμως η απλούστευση να βοηθήσει για να επιταχύνει την εφαρμογή επιτόπου των πολιτικών. Αυτή είναι η, ο διπλός στόχος, η διπλή επιθυμία. Και σε αυτό το πλαίσιο κάναμε την πρόταση απλούστευσης και την έχουμε συνοδεύσει με δύο άλλες προτάσεις που θα τις συζητήσω. Ε, βασικά λοιπόν, απλούστευση. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτή για τα βασικά προγράμματα. Γιατί πολλά χρήματα δαπανώνται μέσω των μεγάλων προγραμμάτων. Τι έχουμε απλουστεύσει καταρχάς σε πρώτη φάση. Υπάρχει μόνο ένα κατόφλι 50 εκατομμυρίων ευρώ για όλα τα μεγάλα προγράμματα στο μέλλον. Ενώ μέχρι σήμερα είχαμε δύο. Ένα 25 εκατομμύρια για τα περιβαλλοντικά προγράμματα και ένα 50 εκατομμύρια για τα υπόλοιπα προγράμματα. Και υπήρχε το πρόσθετο πρόβλημα ότι με βάση, ανάλογα με το ταμείο, ε, ταμείο συνοχής κτλ. ή άλλο ταμείο, το τι είναι περιβαλλοντικό πρόγραμμα και το τι είναι μη περιβαλλοντικό ορίζεται με διαφορετικούς ε, τρόπους. Επομένως, βάλαμε ένα κατόφλι, έναν ορισμό και έχω την εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτό το μονοδικό κατόφλι είναι πραγματική απλούστευση και μειώνει και τις συγχύσεις και τα προβλήματα. Δεύτερον, έχουμε απλουστεύσει τη διαχείριση των μεγάλων προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προγράμματα εθνικού, εθνικής εμβέλειας ή κοινοτικής εμβέλειας αν παραδείγματο χάρη φτιάξουμε ε, μια σιδηροδρομική γραμμή ή έναν αυτοκινητόδρομο που περνάει από πολλέ περιφέρειες, μπορεί να παρουσιαστεί ω ένα πρόγραμμα, ακόμα και αν διατρέχει διάφορες χώρες. Μέχρι στιγμή δεν ήταν δυνατό αυτό και με βάση την εμπειρία μα ε, δημιούργησε τεχνητά προβλήματα, τεχνητές περιπλοκές. Νομίζω ότι είναι λογικό και εφόσον ε, είναι λογικό θα πρέπει να εφαρμοστεί. Επίσης έχουμε αυξήσει την ευελιξία για τα μεγάλα προγράμματα για να συμμορφώνονται με τον αυτόματο κανόνα. Οι εξαιρέσεις που υπάρχουν για τα μεγάλα προγράμματα θα ισχύουν μόνο αυτή τη στιγμή υιοθετηθεί από την Κομισιόν ένα μεγάλο πρόγραμμα. Στο μέλλον αυτός ο κανόνας εξαίρεσης μπορεί να ισχύσει ήδη από την πρώτη στιγμή που υποβάλλεται στην Κομισιόν το πρόγραμμα. Γιατί, Γιατί είδαμε ότι υπάρχουν πολλές, πολλές περιπτώσεις όπου τα προγράμματα είναι τόσο περίπλοκα που χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο από τους τρεις μήνες που προβλέπονται συνήθως για να εγκρίνουμε το πρόγραμμα σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, οι εξαιρέσεις αυτές δεν ίσχυαν, ε, ενώ στο μέλλον θα ισχύουν. Και αυτό νομίζω θα ανακουφίσει τα κράτη-μέλη και θα τα βοηθήσει να επιταχύνουν και από πλευρά του την ε, υποβολή μεγάλων προγραμμάτων. Μοιάζει τεχνικό αυτό, αλλά στην πραγματικότητα σημαίνει ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των προγραμμάτων. Επίσης έχουμε προτείνουμε να πλουστεύσουμε την, τους κανόνες για την αναθεώρηση των προγραμμάτων. Τώρα, περί τι πρόκειται εδώ. Όταν έχετε προγράμματα όπου εισάγονται αλλαγές, τροποποίησεις, ίσονος σημασία στην πραγματικότητα. Συνήθως όμως η εξαίρεση ε, ενός προγράμματος είναι επιλέξιμη όταν υιοθετηθεί το πρόγραμμα. Με βάση τους σημερινούς κανόνες, όταν μετά τροποποιήσεις αργότερα το πρόγραμμα, κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο. Ειδικά σε περίοδους κρίσης θα πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Όταν θες λοιπόν να τροποποιήσεις ε, το πρόγραμμά σου, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να Ό,τι είχε κάνει και ό,τι κάνεις χρειάζεται εκτεταμένη αξιολόγηση. Και ο λόγος που γινόταν ήταν απλό. Ήταν απλός. Σε περίοδους κρίσης δεν χρειαζόμαστε ε, εκτεταμένη αξιολόγηση για να δικαιολογήσουμε την εισαγωγή μιας αλλαγής, ειδικά σε περίοδους κρίσης. Όταν υπάρχουν απειροελάχιστε αλλαγές σε ένα πρόγραμμα, κάτι που μου ήρθε στο, μυαλό για τη Λιθουανία. Έχουμε ένα στάδιο που είχε προβλεφθεί αρχικά για 10.000 ε, θεατές. Και εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια των εργασιών, γίνεται σαφές ότι 10.000 είναι λίγες θέσεις και 12.000 θα ήταν καλύτερο. Τότε, με βάση τους σημερινούς κανόνες, θα έπρεπε να επιλεγεί εκ νέου το πρόγραμμα, στο μέλλον δεν θα χρειάζεται αυτό. Μόνο οι νέες κατηγορίες των δαπανών εισάγονται. Τότε μόνο ε, κοιτάμε νέες ημερομηνίες επιλεξιμότητας. Επίσης προτείνουμε να πλουστεύσουμε τους ε, κανόνες μηχανικής και να τους εφαρμόσουμε κυρίως με σκοπό να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να προωθήσουμε τις ανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάτι πολύ σημαντικό για μας, γιατί θεωρούμε ότι στον τομέα της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, ειδικά σε περίοδους κρίσης, όπως η σημερινή. Και πολλές από αυτές τις δραστηριότητες δημιουργούν και θέσεις απασχόλησης. Επίσης προτείναμε να διευκρινίσουμε διάφορους κανόνες που προκαλούσαν σύγχυση μεταξύ των περιφερειών και ημών. Παραδείγματο χάρη, ένα κλασικό τέτοιο κανόνα ήταν όταν γίνεται μια επένδυση, θα πρέπει να μην ε, γίνονται μετεγκαταστάσεις. Παραδείγματο χάρη, παίρνω από εδώ μια επιδότηση και παίρνω από εκεί, από αλλού μια επιδότηση και φεύγω. Γι' αυτό έχουμε ε, εισαγάγει κάποιες περιόδους ε, για να γίνουν πραγματικές επενδύσεις. Ε, έχουμε εισαγάγει λοιπόν κάποιες περιόδους δέσμευσης, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Επίσης υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες δικτύωσης, δραστηριότητες κατάρτισης. Αυτοί οι κανόνες λοιπόν για τη, οι δεσμευτική. μας μπέρδευαν. Έχουμε διευκρινίσει ότι ισχύουν λοιπόν σε προγράμματα υποδομών και σε παραγωγικές επενδύσεις. Και στην ειδική περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που μιλάει πολύ για κατάρτιση και έχουν πολλά προγράμματα κατάρτιση. Αυτοί οι κανόνες, ε, οι δεσμευτικοί, προβλέπονται υποχρεωτικά από τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με βάση τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Επίσης, σε περίοδους κρίσης, επειδή ζούμε τέτοιες περίοδους, δεν θα εφαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες σε περίπτωση μη κακόβουλων πτωχεύσεων. Κάτι που συμβαίνει με πολλές μικρομεσαίες ειδικά επιχειρήσεις. Υπάρχουν και άλλα μέτρα πλούστευσης που αφορούν την, την παρακολούθηση των εσόδων σε προγράμματα που γεννούν έσοδα λέμε θα το κάνουμε στην επόμενη περίοδο την παρακολούθηση μέχρι το τέλος της περίοδου προγραμματισμού, αλλά όταν συνεχιστεί, όταν τελειώσει ε, η περίοδος προγραμματισμού, δεν θα συνεχίσουμε την, ε, το monitoring, την παρακολούθηση. Κάτι που ήταν μεγάλη ανακούφιση για τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Και έχουμε απλουστεύσει τους κανόνες λογοδοσίας που σε ορισμένες περιφέρειες θεωρούνταν μεγάλο άχθος και έχουμε διευκρινίσει τις εγγύησεις που ζητάμε για να δοθούν προκαταβολές. Ε, για τις κρατικές εγγύησεις ή για τις δημόσιες εγγύησεις που δεν προέρχονται από τράπεζες, έχουμε διευκρινίσει ότι στο μέλλον αυτά, αυτές είναι δυνατές. Επίσης έχουμε δύο προτάσεις που εκφεύγουν λιγάκι αυτού του πακέτου απλούστευσης. Η μία συνδέεται με την κρίση και η άλλη συνδέεται με μια αποτυχία που ανακαλύψαμε. Σας το λέω ειλικρινά στους κανόνες μας. Η πρώτη αφορά την, ε, που αφορά την κρίση είναι η πρόταση στο πακέτο μας για τα χρόνια 2009 να έχουμε μια επιστροφή 100% για τα προγράμματα ESF, του, κοινωνικού, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δηλαδή. Θα είμαι ξεκάθαρο. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε άρδιν τους κανόνες συγχρηματοδότησης. Η επιστροφή 100% για τα έτη 2009 και 2010 δεν θα αμφισβητήσουν σε καμία περίπτωση τις υποχρεώσεις συγχρηματοδότησης που υπάρχουν για κάθε πρόγραμμα. Απλώς σκοπεύουμε το 2009-2010 να δώσουμε την ευκαιρία στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες κάποιες προκαταβολές ε, για να έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες. Μετά όμω, μετά το τέλος αυτής της περίοδου, 2009-2010, θα πρέπει να υπάρξει έτσι μια αποκατάσταση της ισορροπίας για να φτάσουμε στο σύνηθες επίπεδο συγχρηματοδότησης. Δίνω έμφαση εδώ. Το τονίζω, γιατί για αυτό το σημείο νομίζω ότι υπήρξαν πολλές παρεξηγήσεις. Είναι λοιπόν μια πρόταση που η Κομισιόν είχε ήδη αναφέρει στην ανακοίνωσή της για τις κοινέ δεσμεύσει και βρίσκεται για την απασχόληση ιδίω και σε πρώτη φάση επικεντρωνόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Γιατί εδώ όταν υπάρχει αύξηση της ανεργίας πρέπει κάπως να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με γρήγορες δράσεις στα κράτη-μέλη. Τώρα, τελευταίο σχόλιο, Πρόεδρε. Επιπροσθέτως, προτείνουμε μια τροποποίηση του κανονισμού για το Περιφερειακό Ταμείο, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για να καλύψουμε ένα κενό που υπήρχε στο παρελθόν και αφορά την ε, επιλεξιμότητα των ε, παρεμβάσεων για τη στέγαση σε, ε, για κοινότητες έτσι περιθωριοποιημένες, όπως η κοινότητα των Ρώμα και περιορίζεται στις 12 νέες χώρες. Αυτή η πρόταση ανταποκρίνεται σε πολλά αιτήματα που είχαμε λάβει από το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι συνάδει και με τη δική μας ανάλυση. Θεωρούσαμε ότι οι κανόνες που είχαμε ε, για τη στέγαση που συνδέονταν κυρίως με κατοικίες σε αστικές περιοχές δεν ήταν πραγματικά αποτελεσματική. Ειδικά σε ό,τι αφορά αυτές τις περιθωριοποιημένες κοινότητες των Τζικάνων, ας πούμε, που συχνά στην Ήπεθρο και όχι στις πόλεις. Αγαπητοί βουλευτές, αυτές είναι οι βασικές προτάσεις που έχουμε υποβάλει. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει από χθε το Συμβούλιο. Νομίζω ότι ακούστηκε ένας πρώτος γύρος έτσι, σχολείων από τα κράτη-μέλη, κάποιες πρώτες αντιδράσεις. Εγώ προσωπικά δεν μπόρεσα να πάω στο Συμβούλιο χθες, αλλά οι συνάδελφοί μου που ήταν παρόντες μου είπαν ότι σε ό,τι αφορά το πακέτο απλούστευσης, το περιμέναμε ότι θα έχουμε σχετικά θετικές αντιδράσεις, για να μην πω θετικές αντιδράσεις στο Συμβούλιο. Και υπάρχει μάλιστα η βούληση στο Συμβούλιο να πάμε και παραπέρα. Αλλά σε ό,τι σας είπα, αλλά σε ό,τι αφορά το ποσοστό συγχρηματοδότησης κατά 100% ε, για το κοινωνικό ταμείο, εκεί είχαμε αντιρρήσεις στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι θα το συζητήσατε σήμερα το πρωί με την Προεδρία, με την εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Ή θα το συζητήσετε αν δεν το συζητήσατε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στις 11 Σεπτεμβρίου έχουμε μια άλλη συνάντηση στο Συμβούλιο, όχι στις 9 διορθώνει ο μιλτής. Και εκεί θα επικεντρωθούμε στο πακέτο απλούστευσης και καθώς και τις αλλαγές αυτές ε, στο, στον κανονισμό του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τους Ρώμα. Και εκεί υπήρχαν ε, διαφορές απόψεων στο Συμβούλιο. Για τα υπόλοιπα θέματα, στις 11 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα κάνουν ένα τριμερή διάλογο για να συζητήσουν τα υπόλοιπα θέματα, πέραν των άλλων θα συζητηθούν σε 9. Και φυσικά έχω και την επόμενη εβδομάδα ε, μια συνάντηση με το συνάδελφο από την Κομισιόν που είναι υπεύθυνο για το Κοινωνικό Ταμείο την επόμενη εβδομάδα. Και ελπίζω στις 21 Σεπτεμβρίου τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν. δεν φαντάζομαι ούτε κατά διάνοια ότι δεν θα βρεθεί αποδεκτή λύση στο πρόβλημα. Και ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι διτό. Καταρχάς είναι η ρευστότητα στα κράτη-μέλη, τουλάχιστον σε κάποια κράτη-μέλη, που πραγματικά έχουν στεγνώσει από ρευστό λόγω κρίση. Και υπάρχει και ένα ερώτημα που τέθηκε στο Συμβούλιο ε, που δεν υπάρχει στις προτάσεις μας. Ε, το ερώτημα ήταν το εξή από το Συμβούλιο. Ο κανόνας νη συν 2, νη συν 3 του decommitting θα εξακολουθήσει να ισχύει ή θα πρέπει να εξετάσουμε διαφορετικές λύσεις. Αυτά συζητήσαμε. Ελπίζω να μην κολλήσουμε σε αυτά τα πράγματα στους κανόνες, δηλαδή και να κολλήσει ε, η απλούστευση αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε πρόοδο στο Συμβούλιο. Εμπιστεύομαι την Προεδρία. Ενώ τα πιο πολιτικά θέματα που συνδέονται με τη ρευστότητα και τη συγχρηματοδότηση και εδώ μπορούμε να προοδεύσουμε. Αυτά. Ελπίζω ότι θα δουλέψουμε πολύ καλά μαζί πάνω σε αυτό το πακέτο, αλλά θα δουλέψουμε και πολύ καλά για τα υπόλοιπα θέματα που είναι οι προτάσεις ε, για την περίοδο μετά το 2013, καθώς και το θέμα της αναθεώρησης του προϋπολογισμού. Και προς τα πού θα πάει στο μέλλον η Πολιτική συνοχής. Για όλα αυτά τα θέματα ελπίζω να συνεργαστούμε. Είναι δύσκολα θέματα, αλλά πραγματικά μας έχουν συναρπάσει. Εμεί ευχαριστούμε κυρία Νέα και για τους συναδέλφους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα θέματα. Έχουμε συναπόφαση όσον αφορά τον κανονισμό του Ταμείου Περιφερειακή ανάπτυξη και έχουμε αυτό το, αυτή την τροποποίηση για τους ε, Ρωμά, τους Τσιγκάνους. Όλα τα άλλα θέματα θα κρεθούν βάσει τη άλλη διαδικασία, δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη που απαιτείται από πλευρά του Κοινοβουλίου. Και τώρα ξεκινούμε τη συζήτηση. Πρώτος ο Γιάνν Όλμπρεχτ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Γενικέ. Ωραία, ευτυχώς μπορούμε λίγο να δουλέψουμε εκτός της επίσημης κλασικής διαδικασίας δεν έχουμε ακόμα το κείμενο, κατά κάποιο τρόπο προσπαθούμε να προκαταλάβουμε τις εξελίξεις και έτσι βλέπουμε πώς η καλή παράδοση συνεργασία συνεχίζεται. Αν θα αντικαθίσω τον κύριο Φανίστερο που έχει αναλάβει το θέμα για τις διατάξεις αυτές για το κείμενο αυτό έχω να σας πω ένα, μια παρατήρησή μου ότι δηλαδή τώρα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επικρίσεις του ελεγκτικού συνεδρίου προς την Κομισιόν για τον αριθμό των λαθών που έχουν γίνει. Δηλαδή μας λέει ότι θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές διαδικασίες, να είναι πιο καλός ο έλεγχος. Αυτό σημαίνει ότι στενεύουν τα περιθώρια. Περισσότερο από ότι τώρα θα στενέψουν. Από την άλλη μεριά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Άρα, είναι στριμωγμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί θα πρέπει να συγκεράσει αυτά τα δύο πράγματα που απαιτούνται. Από τη μία να είναι πιο αυστηρή, από την άλλη να είναι πιο ευέλικτη. Αυτό το συζητάει και η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και πρώτα απ' όλα κοιτάει το κατά πόσο είναι επιλέξιμε κάποιε δαπάνε. Δηλαδή, εάν κάτι περνάει σε εθνικό επίπεδο και σε ενωσιακό επίπεδο για να αποφύγουμε τις αντιφάσεις. Άρα, εδώ υπάρχουν δυσκολίε. Τώρα ένα δεύτερο στοιχείο. Εδώ συζητάμε και την αυριανή πολιτική. Δεν μπορούμε να πούμε ότι να, σήμερα έχουμε κρίση, να είμαστε πιο ευέλικτοι και σε, σε ένα-δύο χρόνια να ξαναρχίσουμε από το Α και να πούμε α το κάνουμε αλλιώ. Επομένω, αυτό το οποίο εσεί τώρα μα προτείνετε είναι εν μέρη αλλαγή του του συστήματο. δηλαδή να το κάνουμε πιο ανοιχτό, πιο ευέλικτο και να υπάρχει ευθύνη, υπευθυνότητα εκ μέρου των κρατών μελών και εκ μέρου των αποδεκτών αυτών των πόρων. Αυτή είναι υπεύθυνη για αυτά τα χρήματα, για τα προγράμματα. Να η αλλαγή θα γίνει επομένω το σύστημα ευκολότερο, αλλά θα του πούμε, να, εσεί τροφέτε την ευθύνη, αν καταλαβαίνω κατά το πνεύμα που σα διαπνέει. Βέβαια. Τι θα πούν τα κράτη-μέλη. Να έχουν περισσότερο έλεγχο, να έχουν περισσότερη ευθύνη στα χέρια τους και ταυτόχρονα να έχουμε ευελιξία και να είναι τα κράτη-μέλη αποδέκτες των επικρίσεων. Για πέστε μας τώρα κύριε Γενική, είναι δυνατόν να ε, μας μιλήσετε κάπως λιγότερο διπλωματικά. Ξέρουμε κάποιοι μας ότι έχετε κάποιες δυσκολίες με αυτό το πακέτο στο Συμβούλιο. Και περιμένουμε το τελικό κείμενο. Ξέρουμε το βασικό πρόβλημα θα είναι με το κοινωνικό ταμείο ακόμα και αν δεν ανατρέπει όλο το οικοδόμημα. Γιατί σε δύο χρόνια θα υπάρχουν θέματα. Μια που τα ε, κρατημέλη θα πρέπει να πληρώσουν παραπάνω χρήματα μετά το 2010. Δηλαδή, θα εκταμιεύονται πιο εύκολα τα χρήματα, αλλά το σύστημα δεν θα είναι πιο εύκολο. Για πετε μας, πώς βλέπετε τώρα εσείς αυτέ τι δυσκολίε. Για πέστε μας. Είναι δυνατόν να παρακάμψουμε αυτά τα εμπόδια. Τι μπορείτε να μας πείτε τώρα. Εντάξει, δεν θέλω να σας ε, πιέσω τόσο πολύ. Και στα καθήκοντά σας καλή επιτυχία, τι να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταυρακάκης. Thank you, Mrs. Chairman. General. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Γενική Καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξεκίνησε αυτή τη μακρά αλλά και αναγκαία διαδικασία της απλοποίησης. Πιστεύω ότι όλοι στην αίθουσα υποστηρίζουμε τη διαδικασία αυτή. Η πρόταση αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά και ελπίζω να αυξήσει περτέρω τη νομική βεβαιότητα στα κράτη-μέλη και να οδηγήσει τελικά στην πιο γρήγορη απορρόφηση των ε, πόρων. Η πλειονότητα των αλλαγών που εισήχθησαν είναι πραγματικά κατεπίγουσες και ευπρόσδεκτες, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινή διαχείριση των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Αναφέρεται διάφορα θέματα, μεταξύ άλλων το απλό κατόφλι για τα μεγάλα πρόγραμμα, προγράμματα, τους σχετικούς κανόνες, την ενθάρρυνση των έργων που θα οδηγήσουν στην χρήση πράσινων ενεργειών σε ό,τι αφορά την ευελιξία επίσης για την εφαρμογή των κανόνων και σε ό,τι αφορά την κατασκευή κατοικιών για κοινότητες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό, όπως η Ρωμά. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όμως, σε ό,τι αφορά την αλλαγή της 100%, της Και επιτρέψτε μου και κάποιες ερωτήσεις. Ένα από τα βασικά προβλήματα στις χώρες οι οποίες ε, χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση είναι η ρευστότητα. Δηλαδή η διαθεσιμότητα ίδιων πόρων για τέτοια προγράμματα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνειδητοποιήσει ότι υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Με ανησυχεί η λύση της 100% συγκριματοβότησης για το ESF, γιατί καλύπτεται μόνο ένα ταμείο, το οποίο είναι το μικρότερο από τα διευθυντικά ταμεία σε αριθμητικά μεγέθη. Επίσης, ε, το κοινωνικό ταμείο λύνει ένα τμήμα μόνο του προβλήματος της ε, οικονομικής κατάπτωσης. Εκ παραλλήλου, γνωρίζουμε ότι δεν δεν θα υπάρχουν θέσεις εργασίας ακόμα και μετά από την κατάρτιση. Και η τρέχουσα προτάση ενισχύει ουσιαστικά πιο πολύ τα πλέον ισχυρά κράτη-μέλη, ενώ τα πλέον ασθενή λαμβάνουν μόνο 15 επιπρόσθετα ταμεία. Πιστεύετε ότι αυτή η πρόταση είναι η πλέον ε, σκόπιμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευγένη Κυρίλοφ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι μετά από καιρό συζητήσεων χαίρομαι που έχουμε πραγματικά ε, πιέσει προς την κατεύθυνση της απλοποίησης. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες του κυρίου Όλμπριχτ αναφορικά με το ελεκτικό συνέδριο, αλλά εν γέννη η φιλοσοφία θα πρέπει να είναι η εξή. Καλύτερη και πιο απλή. Κανόνες για περισσότερη διαφάνεια για τους ελεγκτές. Συμφωνώ επίσης ότι το τρίτο πακέτο αυτό το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να είναι το τελευταίο, γιατί βρισκόμαστε περίπου στα μέσα της ε, περίοδου αυτή. Γιατί δεν επιταχύναμε την όλη διαδικασία νωρίτερα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι απλό για όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά συμφωνούμε και με την άλλη φιλοσοφία. Ότι οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, πέρα από τις αρνητικές συνέπειες, έχουν και κάποιες θετικές συνέπειες. Ασκούν πίεση, αν θέλετε, για να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και είμαι πεπισμένος ότι οι κανόνες ήταν πραγματικά τόσο περίπλοκοι σε κάποιους τομείς που κάποιοι δικαιούχοι εκ των προτέρων αρνούταν να συμμετάσχουν. Το οποίο ήταν μεγάλο κρίμα ασφαλώ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να καλωσορίσουμε το νέο πακέτο αυτό προκειμένου να καταστεί επικοδομητικό, αποτελεσματικό και να παραγάγει αποτελέσματα το νωρίτερο δυνατό. Να συγχαρώ επίσης τη Γενική Διεύθυνση. Αυτά που συζητήσαμε το Μάρτιο με το προηγούμενο πακέτο, όντως ήδη αποδίδουν καρπούς. Και θυμάμαι ότι είχα εκφράσει κάποιους δισταγμούς τότε. Αλλά είναι καλή η ένδειξη αυτή και με το επόμενο πακέτο νομίζω ότι και πάλι θα πρέπει να καταδείξουμε το ίδιο σθένος προκειμένου να δείξουμε στις χώρες ότι πραγματικά Υπάρχει διαφορά και μάλιστα προτού λήξει η κρίση. γιατί νομίζω ότι υπάρχουν δυσκολίες, αλλά θεωρώ ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να περάσουν το συντομότερο δυνατόν όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση 100% ναι. Θα πρέπει να το συζητήσουμε και να το κοιτάξουμε. Σε γενικές γραμμές όμως, χωρίς να έχω δει το έγγραφο ασφαλώς το λέω αυτό, θεωρώ πάντως ότι θα πρέπει να εκφράσουμε την υποστήριξή μας, την προθυμία μας να επιταχύνουμε τη διαδικασία προς την ε, κατεύθυνση αυτή. Ελπίζω να καταλέξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό και να καταγράψουμε και τη θέση μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αξιότιμη διευθυντά Άνερ. Καταρχάς να σας πω ότι στους φιλελεύθερους είμαστε πεπισμένοι ότι τα μέτρα της απλοποίησης σε κάθε περίπτωση είναι θετικά, αλλά θέλουμε και μακροπρόθεσμα να υπάρχει και μια αξιολόγηση της, ε, του αντικτύπου. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα στην φάση αυτή να επικεντρωθώ σε κάποια ερωτήματα αναφορικά με τη χρηματοδότηση 100%. Γιατί μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε το τι σημαίνουν στην πραγματικότητα οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή ότι θα, θα χρηματοδοτούνται τα κονδύλια 100%, 100% αλλά μετά θα υπάρχει δηλαδή εξισορρόπηση ότι πρόκειται δηλαδή για ένα άτοκο ε, δάνειο προς τα κράτη-μέλη. Και εδώ να ρωτήσω και το εξή. Το πιστοτικό αυτό πλαίσιο είναι απαραίτητο γιατί άλλωστε όλα τα κρατημέλη έχουν προβλήματα πίστοσης. Και όταν μιλάμε για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων σε ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης 20% είναι μικρότερο το ποσοστό συγχρηματοδότησης και υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν προχωράνε τα προγράμματα. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης, μπορεί όμως και επιτόπου να αποφασιστεί ότι όχι, δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε κατά 20% γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Και όταν ε, δίνεται 100% χρηματοδότηση δεν ε, θα υπάρχει ανάλογο κριτικό πνεύμα. Δεν θα εξετάζεται πραγματικά σκοπιμότητα του προγράμματος. Από αυτή την έννοια λοιπόν με απασχολεί το να καταργηθεί η χρηματοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ακριβώς εννοεί αυτό το ποσοστό χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί εκ των υστέρων. Τι εννοείται ακριβώς. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, να απαντήσει ο γενικό διευθυντή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα, για τον Γιάνν Όλμπριχτ. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Αυτές οι απλουστεύσεις που έχουμε εισαγάγει είναι κάποια στοιχεία που θέλουμε να συνεχίσουν να ισχύουν. Και η γενικότερη τάση της πολιτικής μας θα πρέπει να είναι η τάση προς περισσότερη ευελιξία. Και γι' αυτό ισχύει, κύριε Κυρίλοφ, αυτό το οποίο ότι εδώ θα κάνουμε μια πάυση όσον αφορά το πακέτο 2007-2013. Αλλά θα θέλαμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια απλούστευσης και για την περίοδο μετά το 2013. και ελπίζω για την περίοδο εκείνη το 2013 να κάνουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα. Και ελπίζω από την αρχή να τα πάμε καλά, να κάνουμε μια καλή αρχή ούτως ώστε να μπορέσουμε να μεταβάλουμε επιτυχώς τον ισχυρό κανονισμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το πώς θα αποδώσει ο μηχανισμός στο μέλλον. Επίσης, έχουμε συνεχή επαφή με το ελεγκτικό συνέδριο. Μια φορά σωστά ή λάθος μας λένε ότι είναι μπερδεμένη η νομοθεσία που θεσπίζεται και εμείς ελέγχουμε το σύνομο της νομοθεσίας. Κάντε απλούς νόμους μας λένε για να είναι πιο εύκολο και εμείς να ελέγξουμε τις τείχων αντικανονικότητες και τα άλλα που πάσχει η νομοθεσία. Βεβαίω και κάθε φορά είναι αντιχώ και αντιμετώπιση. Όμω τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Είναι πολύ πιο βαθιά τα συστήματα και άρα θα πρέπει και εμεί να κάτσουμε και να δούμε πώ μπορούμε να επιλύσουμε ένα σώρο από κρίσιμα, κρίσιμα θέματα. Ε, να, να σα πω κάτι το, το οποίο το αντιμετώπισα χτε. Δεν το είχα σκεφτεί. Είναι όμω πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Όταν κάποιο εξετάζει το αν υπάρχουν κάποιε αντικανονικότητε που έχουν λάβει χώρα στα κράτη-μέλη όσον αφορά την εκτέλεση τη πολιτική, τότε θα ήθελα να σα πω, κοιτάξτε, δεν πρόκειται για τα, τα, τα ποσά. Πετε μου αν είναι λάθο, γιατί έχουμε ένα 60% το οποίο έχει να κάνει με του διαγωνισμού. Ερωτώ. Ο στόχο, ο σκοπό, η δουλειά τη πολιτική συνοχή είναι αυτός είναι ο χωροφύλακας για το αν διεξάγονται καλά οι διαγωνισμοί. Να, το θέμα ποιο είναι. Και είναι τεράστιο θέμα αυτό. Και δεν είναι δυνατόν με δύο γραμμές να το ξεπετάξει κανείς μέσα σε ένα μικρό έγγραφο. Είναι πολιτικές επιλογές που θα πρέπει να συζητηθούν ακόμα και μετά την περίοδο 2013. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ένα άλλο που θα πρέπει να μας απασχολήσει, ότι θα θέλαμε να κάτσουμε και να φτιάξουμε όλο το σύστημα ελέγχου, να το φτιάξουμε έτσι ούτως ώστε να έχει τα θεμέλια του ε, στις ε, εθνικές διοικήσεις, στις περιφερειακές διοικήσεις και έτσι να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και τι περιφέρειες, δεν ξέρω, α το πούμε συμφωνία κυρίων, συμφωνία εμπιστοσύνη, συμβόλαιο εμπιστοσύνη. Και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μα. γιατί όλε οι ενδείξεις λένε ότι έτσι το σύστημα δουλεύει καλά. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάτσουμε και να του εμπιστευτούμε, μέχρι ότου αποδειχθεί βέβαια το αντίθετο. Ε, εμπιστευτούμε λοιπόν για αλόπιστο ότι τα πράγματα πάνε καλά σε ένα κράτο μέλο. Επίση κάτι άλλο το οποίο δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε έναν κανονισμό που αποσκοπεί σε αναθεώρηση. Πάντως, το θέμα αυτό εγώ το λαμβάνω υπόψη και διαπίστωσα ότι και απασχολεί και εσά σήμερα. Πρόκειται για κάποιε πάρα πολύ πετυχημένε πρωτοβουλίε όσον αφορά τις μελλοντικέ εξελίξεις Κάποιε πρωτοβουλίε αναπτυξιακέ που γίνονται πολλέ φορέ σε τοπικό επίπεδο. Και θα πρέπει και στο μέλλον να κάτσουμε αυτό να το λάβουμε υπόψη και στα πλαίσια τη Εδαφική συνοχή και θα πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθουμε. πώ δηλαδή μπορούμε να κάνουμε περισσότερα ούτω ώστε να βοηθήσουμε σε τοπικό επίπεδο την ε, ανάπτυξη και αυτές τις πρωτοβουλίε πρωτοβουλίες και να εξασφαλίσουμε πώ θα συντεριάζουν αυτές τις πρωτοβουλίες στο γενικότερο ψηφιδωτό της στρατηγικής μας όπως αυτή τη χαράξουμε. Οπότε και οδηγούμεθα στο άλλο θέμα. Αφού πάμε σε τοπικό επίπεδο, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι η διαχείριση θα είναι τέτοια που δεν θα μπλοκάρει τις πρωτοβουλίες. Σας ξαναλέω, είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά για το μέλλον. Επαναλαμβάνω, η τάση, η κατεύθυνσή μας είναι περαιτέρω απλούστευση. Συνεχίζουμε και διαβουλευόμαστε με τους ειδικού που δουλεύουν επί τόπου στα κατημέρια. Θα συνεχίζουμε να συνομιλούμαστε βεβαίω και με εσά, γιατί και εσεί εκπροσωπείτε κάποιε περιφέρειε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε περαιτέρω την κατάσταση. Ναι, τελικά βήμα-βήμα αυτό θα οδηγήσει σε μια αλλαγή του συστήματος. Ε, ε, για τον κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος μας μίλησε για αυτό το 100% της συγχρηματοδότησης για το κοινωνικό ταμείο και με ρώτησε εάν αυτό επαρκεί. Η αλήθεια είναι στο Συμβούλιο υπάρχει μια ομάδα των κρατών μελών που λένε ευχαριστούμε πολύ, αυτό χρειάζεται γιατί έχουμε πρόβλημα ρευστότητος ε, τώρα όμως, όμως το κοινωνικό ταμείο δεν επαρκεί. Δεν είναι αρκετή η τόση όσο χρειαζόμαστε. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Η δε άποψη ότι επικεντρωνόμαστε στο κοινωνικό ταμείο έχει κάποιους, κάποιες αιτίες πρώτα-πρώτα διότι έχουμε λένε και περισσότερα προβλήματα ανεργίας γιατί τα μέτρα του κοινωνικού ταμείου είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα. Τώρα τα μέτρα του Ταμείου Περιφερικής ανάπτυξη. μας οδηγούν σε κάποια βραδίτητα Και δεν είναι η έλλειψη πόρων. Οι λόγοι της βραδίτητα έχουν τι ρίζες τους στην πολυπλοκότητα των μεγάλων προγραμμάτων και αλλού. Πάντως, το ερώτημα παραμένει πώς θα υπάρχει αρκετή ρευστότητα υπέρ των κρατών μελών, ιδίω τα κρατημέρια τα οποία χτυπήθηκαν πιο σκληρά από την κρίση. Και έτσι μένει δυνατόν να αναλυθεί δράση άμεσα. Τώρα. Ήδη έχουμε κάποιε προκαταβολές που έχουν καταβληθεί. Ήδη στο τελευταίο πακέτο αυτές οι προκαταβολές έχουν ε, αυξηθεί. Θα έχουμε παραπάνω ε, 6,5 δις αν θυμάμαι καλά οπότε κανονικά θα πρέπει το μηχάνημα να είναι εντάξει από πλευρά ρευστού ο μηχανισμός σε σχέση με αυτή την πρόταση και αν θέλουμε να έχουμε κάποιο συγκεκριμένο στόχο βέβαια αυτό, αυτό και κάνουμε αλλά ε, όχι όχι δεν, δεν πρόκειται για χρήματα παραπάνω Πρόκειται για κάποια χρήματα που είχαν προβλεφθεί να καλύψουν όλη αυτή την περίοδο και τα οποία είπαμε ότι άρχισαν να τα ευθύ εξ αρχή και μόλι τελειώσει η περίοδο 2000-2010 όλα αυτά τα χρήματα προ το τέλο τη περίοδου θα πρέπει να επιστραφούν. Όταν έχουμε κάποιο πρόγραμμα του Κοινωνικού Ταμείου, κατά τη γνώμη μου, 2009-2010, τότε καταβάλουμε ότι προβλέπει η συγχρηματοδότηση αλλά δίνουμε στο, στο, στο, στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος μία προκαταβολή ένα ποσό παραπάνω που πάμε μέχρι το 2010 τίποτα άλλο όμως παραπάνω τίποτα άλλο δεν προκαταβάλλεται και μιλάμε για τις χρήσεις 2009 και 2010 και αυτό έχει σημασία, πρέπει να το ξέρει το Κοινοβούλιο γιατί είναι αρχή του προπολογισμού, αυτά τα χρήματα εντάσσονται στο σχέδιο του προπολογισμού για τη χρήση 2010. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η προκαταβολή μπορεί να υποστηριχθεί σύμφωνα με όλες τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, τις προβολές, μπορεί να υποστηριχθεί από τον προπολογισμό του 2010 ακριβώς όπως προβλέπει το προσχέδιο του, του, του, του, του προσχέδιο της Κομισιόν το οποίο θα, θα υποβληθεί στην αρχή του προπολογισμού για να το συζητήσετε. Το επόμενο τώρα. Το επόμενο. Θερμές ευχαριστίες προς τον κύριο Κύριλοφ γιατί μας υποστηρίζετε βεβαίως και χρειαζόμαστε να μας ε, στηρίζετε και δεν λέω να μας δώσετε επιταγή λευκό αλλά θα πρέπει ταχύως να διεκπαιρεωθεί και να περάσει αυτό το θέμα οπότε και χρειάζεται να μας βοηθήσετε όπως είπατε και εσείς έχει ξεκινήσει αυτή η διαδρομή και θα θέλαμε η διαδρομή αυτή να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του ενεστώτος έτους. Πάντως, θα πρέπει να το τελευταίο πακέτο. Βέβαια ποτέ μιλές, ποτέ, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει σε κάνα δύο χρόνια, αλλά από δική μας πλευράς και συμφωνούν στα κράτη-μέλη οι εμπειρογνώμονες, πρόκειται για το τελευταίο πακέτο. Πάντω έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε και να επεξεργαζόμαστε το πακέτο για την περίοδο μετά το 2013. Κύριε Τάιρα, εσεί επίσης είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε ότι είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο η απλούστευση, αλλά θα πρέπει κανείς να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της σχετικής πολιτικής. Το είπαμε, το ξαναείπαμε τρεις φορές, όμως θα πρέπει να σκεφτούμε ακριβώς τι εννοούμε. Τι αλλαγέ πρέπει να γίνουν για το 2013. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το πώ είναι δυνατόν να μπορέσουμε να θεσπίσουμε κάποια συστήματα τα οποία μα βοηθούν να κάνουμε μια καλύτερη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των, ε, της πολιτικής μας, των προγραμμάτων μας. Ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλά όσον αφορά ε, για την αξιολόγηση εκ των υστέρων του 2006 Έχουμε εκθέσεις, τρέχουν αυτές οι εκθέσεις, θα δημοσιευτούν και οπωσδήποτε και φυσικά και θα σας ενημερώσουμε και εσάς. Ίσως κατά το τέλος ε, της χρονιάς να μπορούμε να συναντηθούμε για να έχουμε μια γενική άποψη του τοπίου, τι, τι, τι, συμπεράσματα έχουμε για την περιοδο του 2000-2006. Αλλά θα πρέπει επίσης να μπορέσετε να κάνετε και να σκεφτείτε για την τρέχουσα περίοδο και ακόμη περισσότερο για το μέλλον πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερα. Εμείς τώρα επεξεργαζόμαστε τη μεθοδολογία και με μεγάλη μας χαρά να επανέλθουμε σε αυτά που είπε και ο κύριος Γιάνν Αλμπριχτ. Μακάρι να υπάρξει στο μέλλον ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο να μην διακρίνεται από αυτή την αιμονή στα λάθη και στις ε, αντικανονικότητες, αλλά να πρόκειται μια διαδικασία μάθησης. Μάθησης για το τι αποδίδει, τι αποδίδει και τι δεν αποδίδει. Τι δουλεύει καλά και τι δεν δουλεύει. Και αν καταλήξουμε εκεί, τότε, τότε θα κρεμάσω τα παπούτσια μου. Θα αποχωρήσω. Ενδόξως. Σημαίνει ότι έχω κάνει τη δουλειά μου. Όμως, Φυσικά και η δουλειά αυτή είναι πάρα πολύ συναρπαστική. Χαίρομαι πάρα πολύ που θίξατε αυτό το σημείο. Θα επανέλθουμε οπωσδήποτε σε αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Άνερτ, τα στοιχεία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι γενικά στοιχεία τα οποία καλωσορίζουμε. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις αναφορικά με το housing, με τις κατοικίες, αλλά και σε ό,τι αφορά τον ε, κανονισμό το γενικό, σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση κατοικιών. Να κάνω μία παρατήρηση. Νομίζω ότι και στην ε, Δυτική Ευρώπη υπάρχουν κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες για τις οποίες θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, κατάλληλες προσφορές. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να εξετάσετε μήπως το εύρος εφαρμογής θα έπρεπε να επεκταθεί. Και θα σας παρακαλέσω να μην ε, είναι στενή η ερμηνεία των κοινωνικά αποκλεισμένων ε, ομάδων. Τώρα, μία παρατήρηση επί της αρχής για τον γενικό κανονισμό για τον οποίο μαντεύουμε προς το παρόν. Αλλά οι προτάσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά αξίζει να μεταφερθούν και στην επόμενη περίοδο. Ένα παράδειγμα για τα μεγάλα προγράμματα, για παράδειγμα. όλα αυτά είναι πραγματικά στοιχεία που μας βρίσκουν σύμφωνους. Ωστόσο, κάτι που προκαλεί μια δυσαρέσκεια. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα ρευστότητα σε κάποια κρατημέλη. Αλλά να θυμίσω τι ήταν αυτό που έκανε δυνατή την Ευρώπη στην κρίση. Ήταν το σύμφωνο σταθερότητας, οι κανόνες της ίδιας ευθύνης για την παροχή πιστώσεων, δηλαδή τέτοια στοιχεία τα οποία απέθυναν έκκληση στην ευθύνη των ίδιων των πολιτών, των ίδιων των επιχειρήσεων, των ίδιων των κρατών. Και θα ήθελα πραγματικά να πω το είπε και ο Γιάνν Όλμπριχτ, ότι υπάρχει ο κίνδυνος στη μελλοντική αρχή της περιφερειακής ενίσχυσης να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί το θέμα είναι το θέμα αρχής. Όταν το κοινωνικό ταμείο υποστηρίζει 80% των προγραμμάτων αυτών, πραγματικά είναι τεράστιο το ποσοστό αυτό. Είναι τεράστια η προσφορά προς τις περιφέρειες. Αν λοιπόν το πρόβλημα είναι το 20% ίσως τελικά τα προβλήματα να βρίσκονται αλλού. Να φταίει η ίδια η ευθύνη των κρατών μελών των επιχειρήσεων των περιφερειών για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Και αυτό μας ανησυχεί. Άκουσα ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά, αλλά ποιος, θα, ποιος μπορεί να πει πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση στη μελλοντική περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν ότι πραγματικά, πιστεύω ότι πραγματικά είναι σωστή η αρχή του να διατηρηθεί η ίδια ευθύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Μία από τις δυνατότητες αξιολόγησης του πακέτου που έχουμε επιτάπητος, πακέτου για την απλούστευση, θα ήταν να αναλύσουμε πώς το Περιφερειακό Ταμείο και το Κοινωνικό Ταμείο ε, εφαρμόστηκαν μέχρι το 2006. Γιατί η 1η Ιανουαρίου 2009 ε, ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή των προγραμμάτων, για τα δύο αυτά προγράμματα, για όλα τα κράτη-μέλη. Και όμως, όμως δεν ολοκληρώθηκαν όλα τα προγράμματα μέχρι αυτή την ημερομηνία και επομένως δεν έχουν στάλει όλες οι τελικές ε, εκθέσεις. Ε, επομένως θα σταλούν και φέτος, μέσα το 2009 και του χρόνου, μέχρι τον Ιούλιο του 2010. Ε, αυτό ήταν πρόβλημα απλούστευσης. Τελικά έτσι θα λυθεί. Γιατί συχνά ε, τα κράτη-μέλη ε, εγκαλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι φταίει η γραφειοκρατία της. Μήπως μερικές φορές δεν έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα γιατί η τοπική διαχείριση είναι κακή, γιατί τα προγράμματα ήταν κακά. Πρέπει να αναλύσουμε γιατί κάποια από τα προγράμματα καθυστέρησαν και γιατί δεν έφτασαν έγκαιρα οι εκθέσεις. Καλό δεν θα ήταν να τα αναλύσουμε αυτά για να μιλήσουμε για απλούστευση. Ε, να μην γίνει δηλαδή μπέρδεμα. Και ένα δεύτερο, να σας δώσω ένα παράδειγμα για την απλούστευση. Μιλήσαμε λιγάκι για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κατοικιών, την ενεργειακή εξοικονόμηση. Με βάση τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου θα δοθούν χρήματα με βάση ένα πρόγραμμα για να γίνει πιο αποτελεσματική η μόνωση των κατοικιών για να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας, θερμότητας εν προκειμένου. Όμως, λέγεται στο πρόγραμμα ότι για να, υπάρξουν, για να δοθούν τέτοια κονδύλια θα πρέπει ε, να υπάρξει ιδιωτική πρωτοβουλία. Ε, κατά 51% θα πρέπει να βγουν τα χρήματα από την τσέπη του, δηλαδή. Όμως τι γίνεται με τους κατοικού που ζουν σε πολυκατοικίε με 100 διαμερίσματα α πούμε. Θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι αυτοί. Ε, στη δική μου χώρα και σε άλλες νέε χώρες δεν είναι εύκολο να πούμε. Κοιτάξτε, πηγαίνετε στην, ε, στην τράπεζα, βγάλτε λεφτά την τσέπη σα για να συγχρηματοδοτηθείτε από την Ευρώπη. Τι θα σας πούνε αυτοί. Ε, μπορεί να πληρώσουμε τώρα, να αυξηθούν οι τιμές ενέργειας και σε τελική ανάλυση να μην κερδίσουμε. Δηλαδή, σε περίοδους κρίσης όπου ο κόσμος δεν έχει χρήματα στην τσέπη, θα ήταν καλό να απλουστεύσουμε τα πράγματα, ούτω ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια για νοσοκομεία, για σχολεία κτλ. Επειδή δεν κάναμε την απλούστευση αυτή, ε, γι' αυτό έχουν κολλήσει κάποια από τα προγράμματα σε ορισμένε χώρες. Ε, θέλω να κάνω μια ερώτηση για την καθυστέρηση της συγχρηματοδότησης. Τι θα γίνει το 2011, 2012, 2013, εάν γίνει κάτι και δεν πληρωθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Και τι θα γίνει σε αυτούς που δεν είναι έτοιμοι για συγχρηματοδότηση. Γιατί ξέρετε καλά, αν υπάρξει καθυστέρηση και αναβληθεί η, συγχρηματοδότηση για το 2012, 2013, 2014 κτλ. Ξέρετε πολύ κάτι συμβαίνει. Αυτά τα δάνεια θα γίνουν κακά δάνεια. Ο κύριος Ματούλα. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, ευχαριστώ. Σας ε, συγχαίρω για το πακέτο μέτρων που σκοπεύουν την απλούστευση. Είμαι πεπισμένος ότι αν εγκριθεί αυτό το πακέτο, εμπρόθεσμα, θα πετύχει τους στόχους του το συντομότερο δυνατό. Θα ήθελα να σας θέσω ένα πρόβλημα μετά από τη συζήτηση που κάναμε στην ομάδα εργασίας. Προτείναμε λοιπόν να αντικαταστήσουμε τον κανόνα νησιν 2 από τον κανόνα νησιν 3. Η Ρουμανία και άλλες ε, χώρες της περιοχής προτείνουν, προτείνουν να γίνει αυτή η αλλαγή γιατί είναι απλούστευση. Αυτή η πρόταση δεν υπάρχει όμως στο κείμενο που μας υπέβαλε το Συμβούλιο. Θα, θα ήθελα να μου δώσετε μια απάντηση. Ευχαριστώ. Κύριος Όρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ την προσοχή στη μεγάλη εξάρτηση των οικονομιών που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα από τις εισαγωγές. Μερικά νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανακοινώσει ένα πρόγραμμα τρομερά φιλόδοξο ε, ενεργειακής αυτονομίας τα επόμενα 20 χρόνια. Παραδείγματος χάρη η Ρεουνιό, όπου βλέπετε συνδυασμένες προσπάθειες της περιφέρειας της Ρεουνιό και του γαλλικού κράτους για να περάσουμε στην ηλιακή ενέργεια, στην αιωλική ενέργεια, στη θερμική ενέργεια και στην έρευνα για την ενέργεια της θάλασσας, τη βιομάζα κτλ. Το ερώτημα που θέτω είναι το εξή. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ποια ιδιαίτερη προσπάθεια μπορούσε να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνοδεύσει αυτές, αυτά τα νησιά που κάνουν μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια. Δεν πρόκειται μόνο για προγράμματα υπάρχουν ήδη απτά αποτελέσματα. Και για να σας συνεχίσω το παράδειγμα της Γρινιό, το 36% της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό το ποσό, το ποσό θα αυξάνει χρόνο με χρόνο αυτό 36%. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλό θα ήταν να κάνει και αυτή μια προσπάθεια για να συνοδεύσει αυτά τα νησιά, όταν ξέρουμε τι διακυβεύεται εδώ στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το, τα διακυβευόμενα δεν αφορούν μόνο την ε, βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών αυτών, αλλά το ίδιο το περιβάλλον. Ε, το κοινωνικό περιβάλλον, δημιουργία θέσεων απασχόληση, ακόμη και την οικονομία ανεξαρτησία των νησιών μας από τις εισαγωγές πετρελαίου, άνθρακα κτλ. Από τα, ορικά από τα ορυκτά καύσιμα εν γέννη. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει μια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει από τα νησιά. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ασύμμορφο με τις ανακοινώσεις που έκανε η Σουηδική Προεδρία προς μια πράσινη οικονομία, προς μια νέα οικονομία. Προηγουμένως ακούσαμε και την κυρία Όλουφσον, την Υπουργό, της Σουηδίας που μας μίλησε πάρα πολύ θετικά για όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σρόντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν παρακολουθήσατε τις πρώτες σας ε, παρατηρήσεις, κυρία Άνερ, αλλά ενημερώθηκα από τους συναδέλφους που κράτησαν σημειώσεις και φυσικά και έχω διαβάσει αναλυτικά το έγγραφο. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να πω ότι συμφωνώ με, ε, το γενικότερο έργο σας, γιατί στο σημείο αυτό χρησιμοποιείτε όλες τις προηγούμενες εμπειρίες σε ό,τι αφορά τα πολιτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα οποία ήταν πολύ, ε, είχαν σταθεί με μεγάλη επιτυχία. Και νομίζω λοιπόν ότι αυτό αποδείχτηκε και στην πράξη, επειδή εξαντλήθηκαν ακριβώς λόγω της επιτυχίας του στα ταμεία αυτά. Θα ήθελα, ωστόσο, στο σημείο αυτό να κάνω και ένα σχόλιο. θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ασφαλείας που Είπατε ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν πιο πολύ σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Υπάρχει επί της αρχής το σύστημα ασφάλειας, το οποίο ενσωματώνεται στην νομοθεσία. Υπάρχει το σύστημα του εταιρικού, του ελέγχου των εταίρων και να ξέρουμε ότι οι εταίροι εκπληρώνουν με σοβαρότητα τον ρόλο τους εκεί που συμμετέχουν και επίσης διαπιστώσαμε στις διασκέψεις ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που πολύ απλά αγνοούν αυτή την αρχή των εταίρων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόλα αυτά προχώρησε τότε στην έγκριση των ε, λειτουργικών προγραμμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να μάθει από τα παθήματά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να φροντίσει σε όλα τα κράτη-μέλη να υπάρχουν πλήρη δικαιώματα για τους εταίρους αυτούς. προκειμένου να εκπληρώνουν και το καθήκον τους, το οποίο περιγράφεται στον κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν έχει κάποιους εταίρους, κάποια άτομα επικοινωνίας, θα πρέπει αυτά τα άτομα να διευκρινίζουν τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά. Αυτό φυσικά μπορεί να ενέχει και κάποιο στοιχείο υποκειμενικής αξιολόγησης, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα κρύβουν τον κόδωνα του κινδύνου και θα εναπόκειται σε εμά να αποφασίσουμε αν θα το εξετάσουμε ή όχι στη συνέχεια. Γιατί η δαλο όπω αναφέρθηκε και από άλλου συναδέλφου, υπάρχει ο κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν τα μία αυτά ω τμήμα του δικού του προπολογισμού, του εθνικού προπολογισμού. Και νομίζω ότι δεν ε, συνεπάγεται επιβάρυνση στα κράτη-μέλη εκείνα όπου τα προγράμματα αυτά ε, δεν παρουσιάζονται ως προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση προβαίνει σε τόσο μεγάλες χρηματοδοτήσεις, αυτό πρέπει σε κάθε περίπτωση πάντα να καθίσταται σαφές προς το κοινό, προς τους πολίτες. Και δεν συμβαίνει αυτό πάντα. Και πρόκειται για θέματα τα οποία έχουν μεγάλη αποδοτικότητα. Και φυσικά το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι ο κόσμος και πιστεύει όταν ένα πρόγραμμα για την απλούστευση, για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζει τους ίδιους τους κανόνες για το περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μα το βλέπει αυτό ο κόσμος. Το διαπιστώνει ο κόσμος. Και είναι πλήγμα για την Ένωση αυτό. Δεν είναι η Ένωση αυτή που υποστηρίζει την ίδια της την πολιτική τους ίδιους της, τους πολίτες. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει μία απλή δυνατότητα άσκησης ελέγχου. Δηλαδή, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χρηματοδοτήση προγραμμάτων τα οποία δεν τηρούν το ευρωπαϊκό περιφερειακό εθνικό δίκαιο και που αντίκειται στα περιβαλλοντικά πρότυπα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει παραβίαση του κινητικού δικαίου και θα πρέπει και να τηρούνται και οι άλλες αρχές του κανονισμού που αναφέρονται στην αρχή σε ό,τι αφορά την διάσταση του φύλου, την κατάργηση των συνόρων και ούτω καθεξής και όλα αυτά δεν νομίζω ότι κοστίζουν πιο πολύ κόπο, χρόνο, χρήμα Απλά θα πρέπει να υπάρχει σωστός προγραμματισμός στους κανονισμούς. Ε, όταν τα απαιτούμε αυτά τα στοιχεία, θα τα λαμβάνουμε και θα πρέπει επανειλημμένα να τα ελέγχουμε για να ενισχύουμε τα προγράμματα αυτά. Και όπου υπάρχει μεγάλη ιδιωτική χρηματοδότηση, είναι ακόμα πιο σημαντική η διάσταση του ελέγχου. Για τα ταμεία λοιπόν αυτά, τα ανακυκλούμενα, νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί. Δεν είναι οι τράπεζες αυτές που ορίζουν τα κριτήρια. Οι, επιτροπές, οι ανάπτυξης είναι αυτές που πρέπει να ορίζουν τους σχετικούς όρους και αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό σας και αυτό πιστεύω ότι θα είναι μοιραίο σφάλμα. Άρα εκεί θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση. Χωρί κόπο, χωρί παραπάνω χρήμα, νομίζω ότι θα ενισχύσουμε του ε, στόχου μας. Σα Σας ευχαριστώ. Αντιδράσει. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Γενικέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. πρώτα απ' όλα, το οποίο είπε και ο Σπίπερ. Ναι. Ήδη ακούσαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Και τα λάβαμε υπόψη. Θα τα συζητήσουμε αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες και θα μπορέσουμε να τα εξετάσουμε και να επανέλθουμε. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για περιθωριακές ομάδες υπερθωριοποιημένες και μιλάμε για τους Ρωμά δεν σημαίνει αυτό ότι κάποιον άλλο τον αφήνουμε απ' έξω γιατί μιλάμε για τον άλλο. Μην έχουμε παρεξηγήσεις ε, για αυτό το θέμα. Γι' αυτό το ποσοστό 100% ναι. Υπάρχει για αυτή τη διετία, είπαμε, η προκαταβολή και κάτι άλλο που ξέχασα να το πω. Πρόκειται για κάτι στη διακριτική ευκαιρία των κράτων μελών. Και ιδίω έχουμε κάποια κατημέρια που έχουν ιδιαίτερε δυσκολίε, όπω α πούμε η Λετωνία. Ίσως ε, προσφέρει και το ενδιαφέρον αυτό το μέτρο, αλλά θα πρέπει τελικά να γίνει απόδοση των χρημάτων. Και αυτό έχει ανακύψει και στο Συμβούλιο από πολλά μέλη. Είναι σε εισαγωγικά θέμα φιλοσοφικό το πώς θα τρέξει το Ταμείο. Τώρα, κύριε Γκότμαν, για την ε, Λετωνία. Με ενδιαφέρει προσωπικά το θέμα. Είμαι σε συνεχή επαφή με τις αρχές της χώρας. Και πασχίζουμε να δούμε πέραν αυτού του κανόνα του 100% τι δυνατές λύσεις να τον εξευρεθούν για τα προβλήματα. Όπως και εσείς τα απαριθμίσατε. Τώρα όσον αφορά την ε, Μόνο στα δημόσια κτίρια και όσον αφορά την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τέτοια δημόσια κτίρια βεβαίω και πάντοτε αυτό μπορεί να τύχει υποστήριξη εκ μέρους μας με τους πόρους της ε, Ένωσης. Κύριε Ματουλέ, έχετε δίκιο, όχι δεν λέει τίποτα η πρόταση όσον αφορά ε, αυτό το οποίο μας αναφέρατε και κατά τη γνώμη μου Ποτέ δεν ήταν τελείως ξεκάθαρο κατά πόσον αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Στην αρχή της χρονιάς θεώρησα ότι το 1 συν 2 θα ήταν ένα τεράστιο θέμα για το 2009. Όμως, από ό,τι μου λέει συνάδελφοι, μετά τις διακοπές είχαμε τόσες πολλές ε, αξιώσεις που τελικά το θέμα θεωρείται περιορισμένο όσον αφορά το 2009. Όμως ίσως το 2010 τα πράγματα είναι πιο σκούρα, πιο δύσκολα. Το είπαν πάντως πολλά κρατημέλη, το ανέφεραν. Άρα αυτό θα πρέπει να συζητηθεί. Και άλλο. Επίσης μας μιλήσατε όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα νησιά. Και ειδικά μας δώσατε το παράδειγμα της Ραϊνιού. Αυτή είναι μια πραγματική ανησυχία που βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας. Νομίζω ότι πολλά νησιά εστιάζουν τις προσπάθειές τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είναι σημαντικό, σημαντικές για το μέλλον τους. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια του σεβασμού των κανόνων μας για να βοηθήσουμε. Τα νησιά αυτά να σας υποστηρίξουμε με σκοπό να υποστηρίξετε και να εφαρμόσετε αυτές τις στρατηγικές στη ΡΕΙΝΙΟΥ. Μην ε, διστάζετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Ε, θα είμαστε στη διάθεσή σας για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ ο Σούλτερ για την ενθάρρυνσή σας, για την πρόταση για το κοινωνικό ταμείο. Συμφωνώ 100% με αυτά που είπατε για την εταιρική σχέση και μίλησατε για τη δουλειά κατοίκων. Χρειάστηκε να κάνω μία ενδοσκόπηση. Πρέπει να κάνουμε ο καθένας τη δουλειά του. Πρέπει να συνεργαστούμε με αλλά πραγματικά είναι στη, στην ατζέντα μας το δεύτερο εξάμεινο να ενδυναμώσουμε τις επαφές μας με διάφορες οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών. Προκειμένου, καταρχάς, να εντοπίσουμε από κοινού πού είναι τα προβλήματα, μαζί τους, έτσι. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τα διορθώσουμε. Και για την περίοδο 2007-2013, αλλά και για να δημιουργήσουμε ένα κανονισμό για την περίοδο μετά το 2013. Ούτως ώστε από το 2013 και μετά πράγματα να ξεκινήσουν με το καλό πόδι. Ε, ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε λάθη και παρατυπίες. Αυτό που λέει το ελεγκτικό συνέδριο. Λάθη και παρατυπίες. Α, όσο μεγαλύτερη διαφάνεια, όσο περισσότερος δημοκρατικός έλεγχος, όσο περισσότερη διαφάνεια στην εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων, τόσο περισσότερες ελπίδες υπάρχουν να εντοπιστούν τα προβλήματα νωρίς και να διορθωθούν. Το σημείωσα το, την υπόδειξή σας, την υπόδειξή σας ό,τι αφορά τα ανανεώσιμα ταμεία και οι οικονομολόγοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, ασχολούνται με τα κριτήρια για τα ανανεώσιμα ταμεία ή τα ανακυκλούμενα ταμεία πώς θα ποια θα είναι τα κριτήρια για να δοθούν τα χρήματα στον τελικό δικαιούχο. Ε, εκεί έχουν και ένα λόγο οι επιτροπές παρακολούθησης. Ο συνάδελφός μου τα σημείωσε και αυτό θα το δούμε τάχιστα. Και αν έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα, σας παρακαλώ να μου τα δίνετε, να μου τα λέτε, γιατί πραγματικά μας βοηθάνε να, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται και να αναλύσουμε τι κρύβεται από πίσω. Τμήμα του προβλήματός μας καμιά φορά είναι ότι τα πράγματα μοιάζουν επί χάρτου 100% καλά, αλλά όταν βλέπεις πώς εφαρμόζονται στην πράξη, έχεις ρίγη. Εδώ όμως χρειαζόμαστε τη δική σας συνεισφορά, τη δική σας συμβολή και εσείς έχετε την απαραίτητη πείρα για να μας βοηθήσετε. Όταν μιλάτε όμως για επαφές με τις οργανώσεις, πραγματικά ομολογώ ότι πρέπει να κάνουμε μια ενδοσκόπηση εμείς στη γενική μας διεύθυνση. Πρόεδρε, αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Στυμπνέρ για την ενδελεχή συζήτηση, την πολύ συγκεκριμένη. Είχα πει από την αρχή, κυρία Γενικέ, ότι κάποια θέματα είναι επίγοντα. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα ξοδέψει το χρόνο ακριβώς που χρειάζεται για να περάσουν αυτά τα κείμενα από τη συναπόφαση. Όχι παραπάνω. Ελπίζω να λάβουμε σύντομα από τους εισηγητές το χρονοδιάγραμμα για την όλη διαδικασία και μόλις έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες ε, αλλά και μόλις έχετε εσείς πληροφορίες ε, για τις συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο θα θέλαμε να αλληλοενημερωθούμε. Από αυτά που ακούσαμε από σας σήμερα, από την Προεδρία σήμερα και χθε, το πρόγραμμα εργασίας της Γενικής σας Διεύθυνσης στους επόμενους μήνες είναι πολύ βαρύ. Ε, πολύ πλούσιο καλύτερα θα έλεγα. Ελπίζω λοιπόν ε, να βλέπω συχνά τους εκπροσώπους σας. Η δέσμευσή σας να μας πείτε ε, ποια ήταν τα αποτελέσματα αξιολόγησης για την προηγούμενη περίοδο είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πολλούς νέους συναδέλφους. Ε, θέλω να το τονίσω αυτό. Και γι' αυτό θα ήθελα να ενημερώνονται για τις επισκέψεις των ε, επιτρόπων στους εκλογείς μας. Θα ήταν χρήσιμο για μας. Κάτι άλλο, κυρία Γκρέλ. Χρειάστηκε να φύγει νωρίς το πρωί. Μας είπε ότι υπάρχει μια ομάδα εργασίας στην ε, γενική σας διεύθυνση για την περίοδο μετά 2013. Ε, από ό,τι φαίνεται όλοι προσωπούνται εκεί, σε αυτή την ομάδα εργασίας, εκτός από εμά. Θα θέλαμε κάπως να εκπροσωπηθούμε και εμείς αυτήν την ομάδα εργασίας. Γιατί είναι χρήσιμη μια διασυνεργασία, χρήσιμο παρακολουθούμε αυτές τις συζητήσεις. Και χρήσιμο για τους Ευρωπαίους τελικά. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, άλλα σχόλια, ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή. Εκτιμούμε την παρουσία σας εδώ. Ξέρω ότι εγώ τουλάχιστον και πολλοί από εμά, ε, ο Γενικό Διευθυντή μόλι γίνεται στο νοσοκομείο. Μέχρι χθε ήταν στο νοσοκομείο ακόμα. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την προσπάθειά σα. Σα παρακαλώ οι υπόλοιποι μείνετε ακόμα για ένα σχόλιο, για ένα σημείο και μετά θα φύγετε.

Τελευταίο σημείο. Ποια είναι η ημερομηνία της επόμενης ε, συνεδρίας. το πράγμα είναι λίγο περίπλοκο. Θα ξέρετε ότι την επόμενη συνάντηση την έχουμε προβλέψει για Δευτέρα και Τρίτη, 5 και 6 Οκτωβρίου. είναι η εβδομάδα των ανοιχτών θυρών στις Βρυξέλλες. Στις 6 Οκτωβρίου στο ημικύκλιο θα έχουμε την έναρξη των ανοιχτών θυρών. 3 με 5 το απόγευμα. Και η συνεδρίαση της Ρέτζη θα είναι αμέσως μετά την έναρξη. Μετά τις 5. Στις 6 Οκτωβρίου το πρωί έχουμε τη συνάντηση της Ρέτζη και μετά έχουμε δύο 2,5 με 4 και 4 μια συνάντηση. Όχι, συγγνώμη, έχει, υπάρχει μια άλλη συνάντηση μια άλλη επιτροπή και μετά εμεί. Αυτά είναι ασυνήθιοι ε, στον προγραμματισμό μας. Θα ενημερώσουμε όμως τους βουλευτές μόλις καθιερώσουμε το πρόγραμμα. Μόλις κανονίσουμε το πρόγραμμα. Κάτι άλλο, δεν ξέρω να σας το στείλω Μιγγέλ. Η Επιτροπή θα οργανώσει συνεδριάσεις για να ενημερώσει όλους τους συναδέλφους για την πολιτική, όσοι, όσοι ενδιαφέρεστε, έτσι. Ε, όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να παρουσιαστείτε σε αυτά τα σεμινάρια. Θα σας ενημερώσω, έτσι, για να είστε παρόντες ε, σε αυτή τη συνάντηση.